Καλώς ήρθατε και πάλι, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, μετά από τις διακοπές που ελπίζω να σας ξεκούρασαν, αλλά υπάρχουν πολλά ανησυχητικά πράγματα στον κόσμο, δεν είναι και ασύνηθες, γιατί ακόμα και στις ε, χριστουγεννιάτικες διακοπές πολλά συμβαίνουν στο πεδίο των ανθρώπινων δικαιωμάτων όταν δεν υπάρχει κανένα εκεί να βλέπει τι γίνεται. Ας Αρχίσουμε λοιπόν την συνεδρίασή μας με την έγκριση της ημερησίας διατάξεως. Ρωτώ εάν ε, μπορούμε να εγκρίνουμε το σχέδιο, το σχέδιο της ημερησίας διατάξεως, αν το εγκρίνετε λοιπόν. Καλό, καλή χρονιά πάλι σε όλους και στους διερμηνείς. Οι διερμηνείς ευχαριστούν και αντέχονται. Και α, νομίζω ότι εγκρίνεται η ημερησία διάταξη, έτσι δεν είναι. Ως συνήθως η συνεδρίασή μας δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και μην λησμονείτε ότι όταν πατάτε το κουμπί του μικροφόνου σας αυτομάτως εστιάζεται η κάμερα στο πρόσωπό σας. Ναι, ναι, έχω μια ανακοίνωση μετά η κυρία Βεροζιά. Όπως είπα έχουμε το λεγόμενο web streaming, σας το υπενθυμίζω, όπου επαναλαμβάνω ότι οι κάμερες, οι τηλεοπτικές κάμερες εστιάζονται στο πρόσωπο σας όταν ε, πατάτε το μικρόφωνο σας, το κουμπί του μικρόφωνο σας. Επίσης να μιλείτε παρακαλώ αργά και καθαρά. Βέβαια εγώ δεν τα καταφέρνω πάντα να μιλώ, καλά, ε, να μιλώ αργά, αλλά ας το κάνουμε για χάρη των διερμηνέων. Ε, ε, ας έχουν υπόψη τους και τα πρόσωπα που κάθονται κοντά στον ομιλητή, στην ομιλήτρια, ότι θα φαίνονται ε, στο διαδίκτυο, ε, με τις κάμερες δηλαδή, και βεβαίως οι υπόλοιποι αστηρούν σιγή. Η κυρία Βερζιά τώρα έχει το λόγο για θέμα διαδικαστικό. Κυρία Πρόεδρε, θα γνωρίζετε ότι από τα μέσα Δεκεμβρίου γίνονται ταραχές στην Τινησία. Δυστυχώς η ε, επιδείνωση ήταν δραματική το Σαββατοκύριακο. Φαίνεται πως υπάρχουν από 20, 30 μέχρι και 50 ε, νεκροί στις τρεις κοινότητες και έχοντας υπόψη και τις συζητήσεις που έχουμε διεξαγάγει παλαιότερα δεν νομίζω ότι μπορούμε να παραλείψουμε σήμερα να αφιερώσουμε χρόνο ε, στο θέμα αυτό. Το θαύμα της Τινησίας αρχίζει και φαίνεται πραγματικά όπως είναι. Ας ε, μην λείψουμε λοιπόν να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Η Πρόεδρος, αρκετές πολιτικές ομάδες έχουν την πρόθεση να ζητήσουν να διεξαχθεί συζήτηση στην, ε, στην ε, περίοδο συνόδου της Ολομέλειας. Ναι, η πολιτική μου ομάδα, λέει η κυρία Βερζιά, θα το πράξει. Νομίζω και η δική σας. Ελπίζω να το κάνουν κι άλλες, γιατί κάπου έχουμε ξεπεράσει τα όρια. Και οι εικόνες που εμφανίζονται παρά την, ε, ε, τους περιορισμούς που επιβάλλει η κυβέρνηση στην Τινησία στο διαδίκτυο είναι πραγματικά αφόρητες. Έχετε απόλυτα δίκιο κύριε Βερζιά. Μπορούμε, μπορώ να προτείνω τώρα αν θέλετε να ε, εγκρίνουμε τα πρακτικά τη συνεδρίαση τη 14η Οκτωβρίου. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις θεωρώ ότι εγκρίνονται. Και έρχομαι τώρα στις ανακοινώσει τη Προέδρου. Δυστυχώ στη διάρκεια των διακοπών πολλά πράγματα συνέβησαν και όχι μόνο ευχάριστα. Θα προσπαθήσω πάντω να είμαι σύντομη. Πρώτα, πριν από την διακοπή των εργασιών μας για τα Χριστούγεννα και το νέο έτος, εγκρίθηκε η έκθεση τη κυρίας και απονεμήθηκε και το βραβείο Ζαχάροφ. Η έκθεση δίνει την βάση στην ε, Επιτροπή μας, χαίρομαι που είναι και η κυρία Αντρικένε εδώ, για να ζητήσει το λόγο από την είπα εκπρόσωπο. Και επίσης λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, η ανακοίνωση για την απόφαση που λάβαμε για βασικούς ορισμούς, διορισμούς μάλλον στην EEAS για τα ανθρώπινα δικαιώματα από την είπατη εκπρόσωπο περιλαμβάνει πολλά από τα στοιχεία που είχαμε ζητήσει να περιληφθούν. Έχουμε και τον Έγγελμπερτ Τόιερμαν που λαμβάνει την θέση του επικεφαλής της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Κοχόμ είναι πρόσωπο πολύ έμπειρο. Ανακοινώθηκε λοιπόν ο διορισμός του λίγο πριν από τα Χριστούγεννα από την ύπατη εκπρόσωπο και Επίσης μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι που η μακρά προσπάθεια που κάναμε να πείσουμε την υπατή εκπρόσωπο να φτιάξει παρατηρητήριο στην, στην εξωτερική, στην υπηρεσία εξωτερικών δράσεων μάλλον, βρήκε θετική ανταπόκριση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, η κυρία Βερόνικα Νόης δεν είναι εδώ, θα έρθει, έχει διοριστεί επικεφαλής της ειδική διεύθυνση Δημοκρατίας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Την κυρία Αγνώτη γνωρίζουμε καλά και έχουμε συνεργαστεί στενά μαζί της. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί σήμερα στην συνεδρίασή μας, αλλά αργότερα. Σας θυμίζω λοιπόν το τι είχε συμβεί πριν από τις διακοπές, όπου το Κοινοβούλιο είχε εγκρίνει έκθεση για το Αφγανιστάν, για την Μαλαισία, εγώ πέρασα μάλιστα τις τελευταίες δυόμιση εβδομάδες στην Μαλαισία, όχι μόνο για να κάνω διακοπές, αλλά και για να, ε, να εξετάσω θέματα ε, φοιτιών φινικελαίου. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Έχουμε μάλιστα καταδικάσει και την πρακτική των ραβδισμών στη Μαλαισία με το ψήφισμά μας. Εγκρίναμε ψήφισμα επίσης για τα θέματα των ομοφιλοφίλων στην Ουγκάντα καθώς και για το δράμα, την τραγωδία των προσφύγων της Ερυτρέα στην έρημο του Σινά. Επίσης, εγώ και ο ε, Έντουαρτ Μακμίλαν Σκότ, αντιπρόεδρος ε, του Κοινοβουλίου Αρμόδιος για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και που είναι απόν αυτή τη στιγμή, βρεθήκαμε στο Όσλο στις 10 Δεκεμβρίου στην ε, τελετή όπου απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στον Λιούξια Ομπο. Ήταν ιδιαίτερα συγκινητική η τελετή αυτή και το ένα, ε, θα έλεγα, αποκορύφωμα της πολιτικής μου σταδιοδρομίας. Ο Έντουαρτ Μακπίλαν Σκότ και εγώ είχαμε την δυνατότητα να ε, ομιλήσουμε σε ένα μεγάλο αριθμό ε, ακτιβιστών από την Κίνα που ασχολούνται με θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων που ζουν όμως εκτός Κίνας δεν μπορούν να επιστρέψουν και οι οποίοι εξέφασαν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες ε, εκπροσωπούνται διπλωματικά στο Όσλο μπόρεσαν να είναι παρούσες. Ωστόσο, 15 έως 20 χώρες αποφάσισαν τέλει να ε, ακολουθήσουν την υπόδειξη της Κίνας να μην συμμετάσχουν στην τελετή απονομής του βραβείου Νομπέλ στον Λιού Ξιαομπό. Κάτι που απασχόλησε όλες και όλους μας πολύ ήταν η κατάσταση στην Λευκορωσία μετά από τις προεδρικές εκλογές που έγιναν στις 19 Δεκεμβρίου. Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ο πρόεδρος Μπούσεκ, ο πρόεδρός μας, ανέλαβε πρωτοβουλία να εγκρίνει έκτακτη συνεδρίαση για την κατάσταση στην Λευκορωσία. Έκτακτη συνεδρίαση που ελπίζω ότι θα συμμετάσχετε όλοι και θα είναι στις 12 Ιανουαρίου, Τετάρτη, μεταξύ μιας 13 ωρών και 15 ωρών. Ε, πρόεδροι των πολιτικών ομάδων επίσης αποφάσισαν να γίνει εξεταστική των πραγμάτων αποστολή στην Λευκορωσία και εξ όσων γνωρίζω πρόκειται να λάβουν τη σχετική απόφαση για την αποστολή αυτή, για τις αρμοδιότητες που, και την εντολή που θα τις δοθούν στις 13 του μηνός. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η απόφαση των αρχηγών ε, πολιτικών ομάδων. Συμφωνήθηκε επίσης ότι η συνεδρίαση της Τετάρτης είναι συνεδρίαση της Επιτροπής ΑΦΕΤ και ε, την συζήτηση διευθύνει ο κ. Αλμπερτίνη, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών ΑΦΕΤ. Θα γίνει όμως σε συντονισμό με την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την Αντιπροσωπεία για τη Λευκορωσία και, και με ε, συμμετοχή της Euronest. Άλλωστε κοινή δήλωση έγινε από τους επικεφαλείς, από τα πρόσωπα που ανέφερα προηγουμένως δηλαδή και δημοσιεύθηκε στις 20 Δεκεμβρίου δήλωση που λέει ότι παρατηρήθηκαν ανομαλίες από τον ΟΑΣΕ στην διάρκεια της ε, διεξαγωγής των εκλογών ότι υπήρξαν επιθέσεις αστυνομικών δυνάμεων κατά διαδηλωτών, ότι αυτά δεν οδηγούν σε επικοδομητικό διάλογο και εκδημοκρατισμό και η σχετική δήλωση του ανακοινωθέν ζητούσε την άμεση απόλυση των κρατουμένων. Ο ίδιος ο πρόεδρος μας κ. Μπούσεκ ζήτησε αργότερα να αποσυρθούν οι κατηγορίες κατά των ε, διαδηλωτών. Και η κοινωνική πλατφόρμα όπως λέγεται, έχει ζητήσει και άλλα πράγματα, ε, δηλαδή μια πλήρη διερεύνηση του τι ακριβώς συνέβη και αυτό είναι σημαντικό. Νομίζω ότι μπορούμε λοιπόν να εκφράσουμε την ευαρέσκειά μας για τις συζητήσεις οι οποίες ξεκινούν σχετικά με τα πιθανά μέτρα που θα ληφθούν εις βάρος των ε, στελεχών της κυβέρνησης της Λευκορωσίας και είναι επίσης σωστό να καταδικάσουμε ε, την ενέργεια της κυβέρνησης της Λευκορωσίας που έκλεισε το γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μίνσκ. Τώρα για το Πακιστάν υπήρξε μια βίαιη δολοφονία του Σαλμάν Ταζίερ, ο οποίος είναι ο κυβερνήτης του Πουντζάμπ και είναι κάποιος ο οποίος έχει γίνει γνωστός για την υποστήριξη που δίδει στις μειονότητες και είναι γενικότερα υπέρ της ανοχής και δολοφονήθηκε από έναν από τους φορούς του. Είχε διαμαρτυρηθεί επίσης για την κακή μεταχείριση ε, του Αζιαν Μπίλ, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο από τα πακιστανικά δικαστήρια για βλασφημία. Ο κύριος Μπούζεκ έχει εκφράσει επανειλημμένα την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απόσυρση και κατάργηση, την πλήρη κατάργηση του ε, νόμου για την βλασφημία που είναι κάτι το εντελώς απαράδεκτο για τη σημερινή εποχή. Υπήρξε επίσης <clears throat> την πρωτοχρονιά και η δολοφονία 21 χριστιανών κοπτών στην Αλεξάνδρεια. Αυτό προκάλεσε διαδηλώσεις των χριστιανών που κατηγόρησαν την κυβέρνηση για την ενθάρρυνση των διακρίσεων εις βάρος τους. Για την ακτή του ελεφαντοστού η κρίση συνεχίζεται, ανησυχούμε ιδιαίτερα. Η Αφρικανική Ένωση έχει ξεκαθαρή άποψη, κάτι το οποίο δεν μας ε, είναι πολύ συνηθισμένο. Και επίσης το ίδιο και η ΕΚΟΒΑΣ, η οποία προσπαθεί να διαιτητεύσει ε, ανάμεσα στους εμπλεκομένους. Παρ' όλα αυτά όμως η υποβόσκουσα παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχίζεται οι αρχές ασφαλείας του Κμπάμπο συνεχίζουν τις απαγωγές και τις δολοφονίες εις βάρος των, οπαδών του Ουαταρά, οι οποίοι και αυτοί βέβαια προβαίνουν συχνά σε βίες ενέργειες. Τώρα στο Σουδάν χθε οι κάτοικοι του νότιου τμήματος ξεκίνησαν την ψηφοφορία στο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία τους. Μέχρι σήμερα δεν είχαμε πάρα πολλά κρούσματα βίας. Θα πρέπει να εκτιμήσουμε τις προσπάθειες και των δύο εμπλεκομένων έτσι ώστε να διατηρηθεί ο ειρηνικός χαρακτήρας. Ο πρόεδρος Μπασίρ λέγει ότι είναι αθώος για τις κατηγορίες εις βάρος του για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου. Εφόσον υπερασπίζεται αυτή την άποψη πρέπει να παρουσιαστεί στο δικαστήριο της Χάγης. Η κυρία Ντοκεζέρ είναι υπεύθυνη της αποστολής μας στο Νότιο Σουδάν και θα παρουσιάσει την έκθεσή της στην επόμενη συνάντησή μας στο τέλος του μηνός Ιανουαρίου όπου θα εξετάσουμε γενικότερα την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Σουδάν. Η κυρία Βερζιά αναφέρθηκε στην Τινησία. Έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για μια αποστολή της υποεπιτροπής μας στην την Ισία. Τέσσερις από εμά θα πάνε εκεί γύρω στις 25-26 Ιανουαρίου. Και εκεί θα προσπαθήσουμε να δούμε με ποιο τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα θίγονται και πώς οι άνθρωποι που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα διώκονται για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε και γιατί υπήρξαν όλες αυτές οι βίες ε, εκδηλώσεις και γεγονότα τις τελευταίες ημέρες. Πρέπει να αναφερθούμε και στην Παλαιστίνη, υπάρχουν πολλά ανησυχητικά συμβάντα, περιλαμβάνονται οι θάνατοι διαμαρτυρωμένων αόπλων πολιτών, έχουν μπλοκαριστεί οι συζητήσεις ειρηνευτικές, Κίνονται προσπάθειες για να ξεκινήσουν πάλι, αλλά δεν έχει υπάρξει πρόοδος. Για την Ουκρανία υπάρχουν κάποιες ανησυχίες. Ήρθα σε επαφή με τον Επίτροπο Φιούλε ζητώντας τον να μου πει μάλλον τι θα κάνει για την επιδρομή των αστυνομικών δυνάμεων σε μια ε, ομάδα κοινωνίας των πολιτών που υπερασπίζεται αυτούς που ζητούν άσυλο στην Ουκρανία. Η ομάδα αυτή ονομάζεται η Νίτσια, η εισβολή της αστυνομίας έγινε στα τέλη Οκτωβρίου και είδα ότι ο κύριος Φιούλε απάντησε αμέσως και με διαβεβαίωσε ότι οι επιτροπές των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσαν το θέμα αυτό με τον πρέσβη εδώ και με την κυβέρνηση της Ουκρανίας και οι εκπρόσωποι των Ουκρανικών αρχών είπαν ότι θα ερευνήσουν την υπόθεση και θα μας ενημερώσουν και εμείς με τη σειρά μας θα σας ενημερώσουμε. Υπάρχουν όμως και κάποια καλά νέα, όχι πολλά δυστυχώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσημα επικύρωσε την σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών με αναπηρίες. Αυτό έγινε στο τέλος του προηγούμενου μήνα η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν τώρα είναι αν θέλετε η πρώτη περιφερειακή οντότητα η οποία υπογράφει μια συνθήκη τέτοιου είδους. Είναι κάτι το οποίο θα ακολουθηθεί από την επικύρωση των μεμονωμένων κρατών μελών όταν δεν έχει ήδη υπάρξει. Τώρα για τη Ρωσία. Ε, έρχομαι στη Ρωσία ιδιαίτερα στα θέματα Χοντορκόφσκι μετά από τις ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν στην τελευταία συνεδρίαση της Υποεπιτροπής θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη ότι όπως ήταν προφανές σε όλους μέχρι τώρα οι ρωσικές αρχές επανήλθαν σε μια κατασταλτική θα έλεγα στάση. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό να βλέπει κανείς ότι η αστυνομία συνέλαβε και κράτησε 150 διαδηλωτές επί τη βάση μιας νομικής ρύθμισης η οποία είναι παράλογη εντελώς. Το είχαμε θέσει το θέμα αυτό μαζί με την κυρία Αντρική και τον κύριο Μπέρμαν. Εν πάση περιπτώσει οι συλλήψεις έγιναν στη Μόσχα αλλά και στην Πετρούπολη και οι κατηγορίες εις βάρος των συλληφθέντων είναι ιδιαίτερα σοβαρές και έχω κάθε λόγο να πιστεύω και ανησυχώ βαθύτατα ότι εδώ έχουμε ε, να κάνουμε με μια μορφή αντίδραση σε κάποια μηνύματα ανοίγματο που έγιναν από τον νέο δήμαρχο της Μόσχας, ο οποίος πιστεύει ότι οι ειρηνικές διαδηλώσεις θα πρέπει να είναι επιτρεπτές. Παρ' όλα αυτά αυτό δεν ισχύει ακόμα και υπάρχουν πολλοί ηγέτες όπως και ο Μπορίς Νεμτσόφ, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, έχει συλληφθεί και αυτός και καταδικάστηκε σε ελαφρά διοικητική κράτηση αλλά εξακολουθεί να είναι ε, στην φυλακή και μου είπαν ότι περνάει πολλές νύχτες σε ένα υπόγειο χωρίς στρώματα, χωρίς κουβέρτες, κοιμάται στο πάτωμα μόνο και μόνο γιατί έχει ε, κάνει κριτική στον Πουτίν τον Πρωθυπουργό. Ελπίζω ο Μπορίς Νεμτσόφ να μπορέσει να βγει και να έρθει να μας παρουσιάσει την κατάσταση στη Ρωσία. Υπάρχουν και άλλα ονόματα, έχουν υπάρξει μάλλον, τα οποία δεν θα αναφέρω τώρα, αλλά είναι απαράδεκτο να κρατούνται ορισμένοι άνθρωποι μόνο και μόνο γιατί ασκούν το δικαίωμά τους για ειρηνική διαδήλωση και για έκφραση ελεύθερης γνώμης. Λοιπόν, θα αφιερώσουμε κάποιο χρόνο επίσης και στην δίκη του Μιχαήλ Χοντορκόφσκι Ενθυμίστε ότι η κυρία Ανδρικίνη, ο κύριος Μπέμαν και εγώ είχαμε εκφραστεί εκ μέρους της Επιτροπής τον Σεπτέμβριο, είχαμε παρακολουθήσει τις διαδικασίες και άλλοι συνάδελφοι επίσης ήταν μάρτυρες της δίκης παλαιότερα. Στις 30 Δεκεμβρίου λοιπόν ο δικαστής Νταβίνκι καταδίκασε το Χοντορκόφσκι ότι έκλεβε πετρέλαιο από την εταιρεία του και προχωρούσε στην έκπληνση των ε, κερδών. Τώρα θα καταδικαστούν προφανώς αυτός και ο βοηθός του μέχρι και το 2017 από ό,τι φαίνεται, αν και θα προχωρήσουν σε έφεση. Ο πρόεδρος Μπούζεκ εξέδωσε μία ανακοίνωση ε, είπε ότι είναι σύμβολο πλέον η περίπτωση Κοντορκόσκη των συστημικών προβλημάτων του κράτους δικαίου και του σεβασμού ή μη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία σήμερα. Βλέπω με μεγάλη χαρά ότι πολλοί από τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει το θέμα αυτό από κοντά είναι παρόντες και θα ήθελα να καλωσορίσω και την κυρία Αλόγκαν η οποία είναι μία από τους υπερασπιστές ε, και νομικούς συμβούλους του κυρίου Χοντορκόφσκη. Για πέντε λεπτά θα σας δώσω το λόγο και θα κάνετε τις παρατηρήσεις που θεωρείτε χρήσιμες ε, για την απόφαση αυτή. Κυρία Λόγκαν, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ah, Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που μου δίνει την ευκαιρία αυτή να ενημερώσω τα μέλη της και τους επισκέπτες εδώ για αυτή την δεύτερη ε, με πολιτικό υπόβαθρο δίκη σε βάρος του Χοντροσκόφσκη και των συνεργατών του. Ευχαριστώ επίσης τους Ευρωβουλευτές για την υποστήριξη που έχουν προσφέρει για την υπόθεσή μας αυτή εδώ και πολλά χρόνια. Ορισμένοι εξ ημών μπορέσατε να παρακολουθήσετε από πρώτο χέρι την δεύτερη αυτή δίκη στην Μόσχα που διήρκεσε πάνω από 20 μήνες. Λίγες πληροφορίες για το ιστορικό της υποθέσεως για όσους δεν γνωρίζετε καλά ε, την υπόθεση αυτή. Το 2003 συνελήφθησαν Χοντορκόφσκι και Λεμπιέντεφ δικάστηκαν για απάτη και φοροδιαφυγή καταδικάστηκαν σε πολιτικού χαρακτήρα δίκη σε ποινή φυλακίσεως 8 ετών το 2005 και το 2007 όταν είχαν ήδη εκτίσει το μισό της ποινή τους τους απευθύνθηκαν νέες κατηγορίες και καθώς αναλάμβανε νέος πρόεδρος στην Ρωσία ο κ. Μετζιέντεφ άρχισε το 2009 πλέον η δεύτερη δίκη πάλι με πολιτικά κίνητρα. Στις 15 Δεκεμβρίου είχε προγραμματιστεί να εκδοθεί απόφαση του δικαστηρίου στην υπόθεση αυτή. Δυστυχώς την ημερομηνία εκείνη, ως γνωρίζετε ορισμένη εξημών, αναβλήθηκε η έκδοση αποφάσεως χωρίς να προβληθούν λόγοι. Εκατοντάδες άνθρωποι περίμεναν στα σκαλιά του δικαστηρίου την απόφαση αυτή. Την επομένη, στις 16, σε τηλεοπτική συνέντευξη του ε, Πρωθυπουργού Πούτιν, που είναι και το ετήσιο διάγγελμά του που απευθύνει στον ρωσικό λαό, του τέθηκε ερώτηση σχετικά με τον κύριο Χοντορκόφσκι, η απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργό Πούτιν στο κοινό ήταν ότι είναι κλέφτης και να μείνει στη φυλακή. Και ότι η δεύτερη υπόθεση Χοντορκόφσκι και Λεμπιέντεφ θα αποδείχθηκε στο δικαστήριο. Και αυτά μία μόλις μέρα μετά την αναβολή της εκδόσης αποφάσεως. Στις 27 Δεκεμβρίου συνήλθε ξανά το δικαστήριο και θεώρησε ότι είναι ένοχος και σκοτωγράφηση για ξέπλυμα χρήματος και απάτη. Κατηγορήθηκαν ότι υπεξήρασαν ολόκληρη παραγωγή, την ολόκληρη παραγωγή του πετρελαίου στη Γιούκος επί έξι έτη. Και τέσσερις μέρες αργότερα, στις 30 Δεκεμβρίου, μόλις μία μέρα ε, πλην, πριν, πριν τον εορτασμό ε, της πρωτοχρονιάς απειγγέλθη η απόφαση. Κύριο Φαντερκόφσκι και ο Λέμπεντερ κατεδικάστηκαν σε 13,5 χρόνια κάθεξε, Δηλαδή μόλις 1,5 χρόνο λιγότερο από την ανωτάτη ποινή που προβλέπεται. Και συνολικά ήταν 14 τα χρόνια σε σχέση με την πρώτη δίκη. Όμως, οι συνήγοροι ακόμα δεν έχουν λάβει την ε, απόφαση. Γιατί είναι αργίες από την 1η Ιανουαρίου στη χώρα. Αύριο είναι πρώτη οπότε αναμένουν την καθρογραμμένη απόφαση μέχρι το Σαββατοκύριακο. Και γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει ε, αυτή η απόφαση ε, ήδη να είχε ε, απαγγελθεί εδώ και χρόνια και να υπάρξει κάποιος συμψηφισμό της κατηγορίας, της ποινή. Οπότε η Χοντροκόφσκι και Λέμπετεφ το 2027 θα απελευθερωθούν οι δε, το δε επιχειρήματα των ε, δικηγόρων τους εγείρουν πολλά ερωτήματα σε σχέση με το πώς θα γίνει η επιμέτρηση της ποινής. Και ρώτησε τους κατηγορουμένους ο δικαστής αν καταλαβαίνουν τις κατηγορίες. Αυτό δεν προέρχεται από τον δικαστή Νίλκιν, αλλά συνεχίζουν και υπάρχουν πολλές εμβολίες από πλευρά των κατηγορουμένων σε σχέση με αυτή τη διαδικασία. Και πάρα πολλές ήταν οι επικρίσεις ε, από τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά αυτή την απόφαση. Ο υψηλό, η υψηλή εκπρόσωπο, η είπατε εκπρόσωπο, η κυρία Άστον, ο κύριο Μπούζεκ, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προέβησαν σε δηλώσει. Ε, ο, ο καγκελάριο τη Γερμανία, η κυρία Μέρκελ, ε, επίση, ε, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, ε, η κυρία Κλίντον, ο Λευκός Σίκος και ε, πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι προέβησαν σε σχετικές επικρίσεις και είναι πάρα πολύ θετικό κατά τη γνώμη μας το ότι στην γενία φωνή από Αμερική και Ευρώπη. Επίσης θα ήθελα σύντομα να σας διαβάσω αυτή τη σύντομη δήλωση των Λιέμπεντεφ και Χοντορκόφσκι κατόπιν της ε, απαγγελίας της ε, ποινής. Και εμείς δείξαμε ότι δεν μπορεί κανείς να υπολογίζει εις την προστασία την δικαστική κατά του κράτους στη Ρωσία. Δεν έχουμε όμως απολέσει την ελπίδα, ούτε εμεί ούτε οι φίλοι μας. Βλέπετε τι θα πει ε, αυτός ο, ο πρώτος νόμος του Τούροφ που είναι ο πρόεδρος της ε, Επιτροπής ε, της Εκλογικής στη Ρωσία και λέει ότι ο Πούτιν πάντοτε έχει δίκιο. Επομένως, ε, άρα, παρόλα αυτά όσα έγιναν, σημαίνει ότι εγώ δεν καταλαβαίνω καλά το τι γίνεται ο νόμος του Τούροφ, λοιπόν. Στις 31 Δεκεμβρίου οι συνήγοροι ε, ίσκησαν κάποιο ένδικο μέσο, κάποια έφεση είναι διαδικασία τρίμηνη έως εξάμηνη ανάλογα με το αν οι αρχές θέλουν να συνεργαστούν ή θέλουν να παρελκύσουν αυτή τη φάση της διαδικασίας. Και πολλέ φορέ ρωτήθηκε ο κόσμο τι θα γίνει με τον Λιαμπεντεφ και τον Χοντερκόφσκι. Θα μείνουν κρατούμενοι στην Μόσχα, πρόκειται να του στείλουν στη Σιβηρία, κάπου αλλού, στη Ρωσία. Και από όσα γνωρίζουμε όσον αφορά τι δηλώσει των σοφρονιστικών αρχών στι 31 Δεκάτου, οι κατηγορούμενοι θα μείνουν εκεί που είναι. Στη, στη, στη φυλακή Ματριόσκα δεν είναι ακριβώς εκεί ένα κάμπινγκ δεν είναι ε, ε, ο, σαν τον τόπο κράτηση τους αρχικά και τέλος πάντων θα μείνουν εκεί μέχρι ότου έρθει η ώρα της έφεσης. Πάντως αυτή δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δικηγόρων τους και των κατηγορουμένων, διότι κατά τις αργίες θεωρείται κλειστή η φυλακή. Άρα, ίσως αύριο θα υπάρξει επαφή με τον κ. Χοντορκόφσκι αν είναι ακόμα εκεί, στη Μόσχα. Thank Εμείς ευχαριστούμε για τη δήλωση που μας ε, διαβάσατε και για όλα όσα μας ενημερώσατε και τώρα θα ήθελα να μιλήσω με τους εκπροσώπους της ε, εξωτερικής υπηρεσίας κύριε Κάρσον για πέστε μας τι, τι πρεσβεύει η υπηρεσία σας όσον αφορά την όλη κατάσταση αλλά και την ε, δικαστική απόφαση έχετε το λόγο σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Οπότε, θυμηθήκαμε τώρα τον background, που, τι προηγήθηκε και πώς έχει κατάσταση σήμερα. Πάρα πολύ θετική μας αυτή η ενημέρωση. Και έχουμε αυτές τις δηλώσεις, έχουμε τις ε, αντιδράσεις οι οποίες προεκλήθησαν, τα όσα είπε η ψηλή εκπρόσωπος στις 31 ε, Δεκεμβρίου, αμέσως μετά την απαγγελία της ποινής. Όπως ε, είπαμε, και εμείς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και οι εκπρόσωποι των κρατών μελών. Ε, βρισκόμαστε όλοι σε συνεργασία ε, όσον αφορά την παρουσία μας στην ε, Μόσχα και υπάρχει συντονισμό μεταξύ των πρεσβειών εκεί αλλά και από πλευράς εξωτερική υπηρεσία παρακολουθούμε τη διαδικασία και σας παραπέμπω στη δήλωση της κυρίας Άστον ότι μας προξενεί απογοήτευση αυτή η απόφαση. Το πώς κατέληξαν τα πράγματα είναι κάτι το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με τις ε, φιλοδοξίες που διατυπώνονται σε ύψιστο επίπεδο ε, ότι δηλαδή πρετανεύει το κράτος δικαίου στη χώρα. Ότι υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και ότι όλοι οι Ρώσοι έχουν το δικαίωμα σε μια δίκαια δίκη. Έχουμε το θέμα της στρατηγικής ε, εταιρικής σχέση με τη Ρωσία και εμείς προσδοκούμε τη Ρωσία να τηρήσει τα όσα έχει υποσχεθεί σε εθνές επίπεδο και συγκεκριμένα τις δεσμεύσει της Ρωσίας στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΗΕ. Αυτά τα είπαμε και τα ξαναείπαμε σε διάφορα βήματα συνεννόησης διαλόγου με τη Ρωσία και πρόσφατα τα είπαμε στις κορυφής Ένωσης Ρωσίας. Του το λέμε και του τα ξαναλέμε. Όπω είπε η κυρία Λόγκεν, είπαμε και τα των δηλώσεων Μπούζεκ και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης επίσης συμφωνεί και χαιρετίζει τις δηλώσεις αυτές. Πρώτη για μια ευκαιρία που είχε η Ρωσία και την έχασε. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία στις 31 Δεκεμβρίου. Επίσης, ε, λαμβάνω σοβαρά υπόψη το ότι ο κύριος Μπούζεκ έθεσε το θέμα της δίκης Χοντροκόφσκη όταν συνάντησε πρόσφατα τον κύριο Μέντεβεντεφ στην Μόσχα. Έχουμε μόνο σε αυτήν την ε, συγκεκριμένη σχέση με τη χώρα. Αυτό ε, ήταν θετικό στα πλαίσια τη συνάντηση κορυφή και θεωρήσαμε ότι υπάρχει δέσμευση για ξενισμό τη οριστική κοινωνία. Αλλά είπαμε ότι αυτό πρέπει να συνοδεύεται και από το κράτο δικαίου. Και εμεί πιστεύουμε ότι ο οικονομικό εξυγχρονισμό δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί χωρί να έχουμε εξυγχρονισμό τη κοινωνία. Οπότε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πριτανεύει το κράτος δικαίου. Τώρα δε έχουμε τα τελευταίες πληροφορίες όσον αφορά το τι αναμένεται να ακολουθήσει όσον αφορά την διαδικασία άσκησης αυτής της έφεσης. Είναι αυτό αυτονόητο όπως παρακολουθήσαμε, θα συνεχίσουμε παρακολουθούμε σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τους άλλους μας εταίρους. και θα συνεχίσουμε προσεκτικά να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Κύριε Κάρσον, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα είπε τι απόψει ο κύριο Κάρσον τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και τώρα ο κύριο Γότσον θα λέει το λόγο που πρόκειται για έναν από του συναδέλφου, ο οποίο ίσω περισσότερο από όλου ασχολήθηκε με τα θέματα τη δίκαιη δίκη, με το τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη δίκη. Κύριε Βότσον, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καταγραφούν στα πρακτικά οι ευχαριστίε μου προ εσά και προ του άλλου συναδέλφου οι οποίοι προσυπέραψαν εκείνη την ε, επιστολή που είχα προωθήσει για τον ε, Πρόεδρο Μέντβεντεφ ε, τον περασμένο μήνα. Όπω γνωρίζετε τώρα δεν πρόκειται για μια αντιπροσωπευτική περίπτωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμω θα γίνει σύντομα περίπτωση παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κ. Χαντροκόφσκι και ο κ. Λέμπεντεφ κατηγορήθηκαν για θέματα εμπορικού δικαίου, θα μπορούσε κανεί να αλλά τελικά, τελικά το έγκλημά του ήταν ότι χρηματοδότησαν κόμματα τη αντιπολίτευση. Όσον αφορά δε όλου εμά που θεωρούμε ότι η Ρωσία είναι ευρωπαϊκή χώρα και που παρά τι δυσκολίε που υπάρχουν ακόμα και θεωρούμε και ελπίζω ότι κάποια μέρα θα μπορέσει. Μου φύγε το τέτοιο. Η τελευταία αυτή καταδίκη και η ανακοίνωση της ποινής είναι ένα σαφές βήμα προς τα πίσω. Στην έκθεσή σας και στην έκθεση της κυρίας Αντρίκεν. Τον περασμένο μήνα είπαμε ποιες είναι οι καθητήρες γραμμές όσον αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπ' αυτές τις συνθήκες. Επίσης ε, καλέσαμε την κυρία Άστον να εξασφαλίσει το ότι ε, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι η ιδέα και το πνεύμα το οποίο θα διαπνέει κάθε, κάθε κίνηση στα πλαίσια της ε, εξωτερικής δράσης. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε αυτά τα οποία γίνονται να μην ε, σχολιάζονται και να μην τα παρακολουθούμε. Η Χριστίνα Όλαντη συνάδελφο, είπε ότι θα πρέπει να προβεί σε κυρώσει. Κυρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ει βάρο τη Ρωσία. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τι λένε οι εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την πρόταση, αυτή την ιδέα. Πάντω και εγώ και άλλοι συνάδελφοι θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαμαρτυρηθεί όσο γίνεται πιο έντονα για αυτά τα οποία συνέβησαν και θα πρέπει να ζητηθεί η απελευθέρωση των καταδικαστέντων και φυλακιστέντων με μέσω αυτής της ε, θλιβερής απογοητευτικής ε, δίκης. Πρόεδρος, ζητήω να το λόγο, δεν βλέπω. Α, εσείς, εσείς. Εσείς κύριε Γκουριάνο, ζητείτε το λόγο. Τον έχετε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ όπως και ο κύριος Βότσον να πω ότι όντως σύντομα αυτή η περίπτωση αυτή η υπόθεση, αυτή η δίκη θα γίνει θέμα παραβίαση των οποίων δικαιωμάτων. Και αποτελεί ακόμα μία συνέχεια στο σύριαλ των σχετικών υποθέσεων στη Ρωσία. Πολιτικόφσκα για Μαγνίτσκι. Έχουν προηγηθεί και άλλε τέτοιε περιπτώσει στη Ρωσία και αν δεν γίνει τίποτα, τότε κάποιο άλλο, κάποια άλλη τέτοια υπόθεση θα ακολουθήσει επίση. Θα ήθελα να πω ότι νιώθω απογοήτευση όσον αφορά την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τώρα για τη δίκη αυτή. Τι κάνει συγκεκριμένα η υπηρεσία εξωτερική δράση για την υπόθεση αυτή. Γιατί τελικά συνεχώς καταλήγουμε στο ίδιο. Στρατηγική εταιρική σχέση με τη Ρωσία που όντως υπάρχει και είναι τέτοια. Αλλά όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, αυτή η εταιρική σχέση και αυτή θα έπρεπε να αποτελεί αφετηρία, πλατφόρμα επικρίσεων. Να είναι ξεκάθαρο και ουσιαστικό το μήνυμα που θα πρέπει να στείλουμε στην Ρωσία. Νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή η νυφάλια, ήρεμη διπλωματία που τώρα κυριαρχεί. Πάρα πολύ σωστά τα είπε ο κύριος Βότσον για τον Χοντροκόφσκι και τον Λέμπιδεφ. Ευχαριστούμε κύριο Σούλς τώρα, ο αντιπρόεδρος της ε, Επιτροπής, ε, της, της Διακοινοβουλικής Επιτροπής σχέσεων με την Τούμα θα λάβει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Εγώ όμως ήθελα να πω ότι δεν έχετε δίκιο κύριε συνάδελφε. Δεν έχουμε τώρα τέτοια στρατηγική εταιρική σχέση με την χώρα. Έχουμε απλώς αυτή την συμφωνία που έχει ως στόχο τον εξυγχρονισμό και ε, το, το θέμα του κράτους του δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι βασικό συστατικό αυτής της συμφωνίας και ε, ο Μέντεβεντεφ και άλλοι ομιλητέ μα είπαν ότι αλλάζουν πράγματα στη Ρωσία. Εγώ δεν συμφωνώ όμω, μάλλον πισωγύρισμα έχουμε παρατηρήσει στην χώρα. Οπότε, φυσικά, τιμήσαμε τον Μαγνίτσι, τώρα όμως έχουμε αυτού που έχουν φυλακιστεί χωρίς αιτιολόγηση και επομένως βλέπετε έχουμε κάποιο είδους νομικιστικό μηδενισμό που πρετανεύδρα στη Ρωσία και κερδίζει συνεχώς έδαφος. Όχι, ακόμα δεν έχει καθαρογραφεί η απόφαση, ούτε δημοσιευθεί. Όμως έχουν τη δήλωση Καζιάνοφ που είπε ότι στην εποχή του δεν θα υπήρχε τέτοιου είδους υπεξαίρεση της παραγωγής πετρελαίου. Πρόεδρος. Κυρία Λόγκεν, έχετε το λόγο. Κυρία Λόγκεν, σύντομο παρακαλώ. Λόγκεν. Δεν έχουμε λάβει ακόμα την γραπτή απόφαση, αλλά από ό,τι λέει ο τύπος και το πρακτορείο Interfax, το δικαστήριο εμήνευσε τη μαρτυρία του Κασιάνοφ ας μη αξιόπιστη. Ευχαριστώ κυρία Λόγκεν. Είμαι βέβαιος ότι η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια και νομίζω ότι όλοι θα υποστηρίξουμε το αίτημα αυτό για περαιτέρω συζήτηση. Να κάνω εδώ μία δήλωση. Δυστυχώς νομίζω ότι υπάρχει μία σύνδεση ανάμεσα σε αυτά τα οποία συνέβησαν με την έκδοση της αποφάσεως Χοντορκόφσκι και Λεμπέντεφ με τα μέτρα που ελήφθησαν εις βάρος των ειρηνικών διαδηλωτών της 31ης Δεκεμβρίου. Να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε επίσης και την αντιπολίτευση της Λευκορωσίας. Γιατί δεν μπορούμε ανοιχτά να υποστηρίξουμε και την δημοκρατική αντιπολίτευση της Ρωσίας. Ξέρουμε ότι έχουμε επαφές και δεν θα πρέπει να δεχθούμε, θα έλεγα, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Υπάρχει και μια ανακοίνωση εδώ η οποία θα σας ενδιαφέρει. Κάναμε προσπάθειες να προσκαλέσουμε τον νέο πρόεδρο της Προεδρικής Ομάδας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να έρθει να μας μιλήσει. Ο κύριος Φέντετοφ προσκλήθηκε να είναι μαζί μας 28 Φεβρουαρίου. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ευκαιρία για μας να ανταλλάξουμε απόψεις για το τι συμβαίνει στη χώρα αυτή ιδιαίτερα με αυτές τις αντιδραστικές κινήσεις οι οποίες γίνονται στην Ρωσία. Μια τελευταία ανακοίνωση. Ο πρέσβης της Σρι με ενημέρωσε ότι υπάρχει ένα κείμενο διαθέσιμο για όλους, το οποίο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή και σχολιάζει τη συνάντηση ε, που έγινε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Σρι Λάνκα μετά την περίοδο της σύραξης. Ξέρω ότι ήσασταν υπεύθυνο κύριε Χάουιτ. Ένα πολύ μικρό σχόλιο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που βοηθήσατε έτσι ώστε να γίνει η συζήτηση για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Να πω επίσης ότι με κάποιο τρόπο στην επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να θέσουμε και το θέμα της επικύρωσης της Σύμβασης των Δικαιωμάτων των Αναπήρων των Ηνωμένων Εθνών είτε στα πλαίσια της ανακοίνωσης του Προέδρου είτε με κάποιο άλλο τρόπο κάτι τέτοιο θα το ιδιαιτέρως χρήσιμο. Νομίζω ότι θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό γιατί οι επικυρώσεις από πλευράς των κρατών μελών δεν είναι κάτι το πάρα πολύ εύκολο και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω το θέμα που αφορά τον πρέσβη του Σιλάνκα και της επιστολής του δεν ήμουν εδώ, αν ήξερα θα προσπαθούσα να είμαι παρόν, αν ήξερα για τη συνάντηση αυτή. Πάντως νομίζω ότι κάθε κυβέρνηση και οι απεσταλμένοι έχουν δικαίωμα απάντησης όταν κατηγορούνται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Του θερήσαμε το δικαίωμα αυτό και είναι πραγματικά λάθος της Επιτροπής μας και θα πρέπει να βρούμε την δυνατότητα να επανορθώσουμε. Δεν ξέρω με ποια μορφή θα το κάνουμε αυτό, ίσως γραπτά να ικανοποιήσει τον αξιότιμο κύριο πρέσβη. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια απάντηση. Ένα άλλο θέμα. Αναφερθήκατε στην ανοιχτή υποστήριξη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Ρωσία και το συγκρίνατε με τη Λευκορωσία. Εγώ δεν είμαι υπέρ της ρωσικής κυβέρνησης, δεν είμαι υποστηρικτής και νομίζω ότι το θέμα της ασυλίας είναι πρόβλημα το θέμα της, ε, με, της ε, ελεγχόμενης δικαιοσύνης είναι πρόβλημα και ε, ο κύριος Κοντορκόφσκι και ο κύριος Λεμπέντεφ έκαναν ό,τι είχαν κάνει πάρα πολύ εκείνη την εποχή και δικάζονται για λόγους καθόλου πολιτικούς. Αλλά η Λευκορωσία δεν είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, δεν σκοπεύει να πάρει μέρος. Η Ρωσία όμως είναι πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και νομίζω λοιπόν ότι αν κάνουμε αυτό το οποίο ζητήσατε θα παραβιάζει το ότι πολλά από τα κόμματα μας έχουν μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, στενές σχέσεις με την ρωσική κυβέρνηση. Το να υποστηρίξουμε λοιπόν την αντιπολίτευση μιας χώρας η οποία είναι πλήρες μέλος της, του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, θα ήταν λάθος. Σέβομαι τι απόψει σα, κύριε Τάνοκ, λέει ο πρόεδρο, αλλά η συζήτηση για τα θέματα αυτά δεν μπορεί να γίνει τώρα. Κύριε Χάουιτ, πολύ σύντομα γιατί ήσασταν προεδρεύων στη συνάντηση για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σρι Λάνκα. Συμφωνώ με την άποψή σας ότι δεν θα πρέπει να γίνει μια τέτοια συζήτηση τώρα. Να πω δύο πράγματα όμως για να μπουν στα πρακτικά να πω ότι σχετικά με τον ε, πρέσβη ε, του Σρι Λάνκα αυτός επέλεξε τη συγκεκριμένη διαδικασία. Δεν είναι αληθές συνεπώς το ότι δεν του δόθηκε το δικαίωμα να πάρει μέρος και να ε, συζητήσει. Δεύτερον, η γραμματεία θα επιβεβαιώσει και ο κύριος Τάνοκ το ξέρει ότι τη απουσία σας ζήτησα από τον Προεδρείο να επανέλθει στο θέμα όχι μόνο ειδικά για τη Σφυλάνκα αλλά γενικότερα στο θέμα αυτό επί της αρχής. Νομίζω ότι με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να ακούσουμε και τις απόψεις των πρέσβεων της Κίνας, του Σουδάν και της Τινησίας είναι θέμα μεθοδολογικό. Θα πρέπει λοιπόν και σε επίπεδο αρχής και μεθοδολογικά να μην περιορίσουμε το πρόβλημα που είναι για συζήτηση στο Σρι στη Σρι Πράγματι θα δούμε ποια είναι η σωστή πρακτική με τους πρέσβεις των χωρών που συζητάμε επανειλημμένα εδώ. Περνάμε στο σημείο 4. Τώρα η ακρόαση για την έκθεση που υιοθέτησε τον προηγούμενο Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ήμουν εισηγήτρια. Δεν χρειάζεται να πω πόσο σημαντικό είναι το θέμα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε σχέση με τις εργασίες μας και σε σχέση με τις εργασίες των υπολείπων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω η έκθεση αυτή να επιτρέψει μια βελτίωση της διοργανικής επικοινωνίας σχετικά με το τι θα πρέπει να κάνουμε συνεργαζόμενοι με την κοινωνία των πολιτών, κάποιοι από τους οποίους είναι παρόντες εδώ σήμερα. σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη πρέπει να φέρουν εις πέρας και να σεβαστούν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει για την υπεράσπιση αυτών που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ήδη από το 2004 και μετά. Πράγματι μια στρεβλή συνέπεια της υιοθέτηση της συνθήκης της Λισαβόνας είναι να είμαστε ουδέτεροι σχετικά με την τύχη των σχέσεων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τα ευρωπαϊκά όργανα. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Σαν παράδειγμα ε, το θέμα των ε, κατεπηγουσών θεωρήσεων έκτακτης, έκτακτης μορφής είναι κάτι το οποίο είναι στα χέρια του Συμβουλίου και πρέπει ε, να τεθεί λοιπόν το θέμα αυτό προς συζήτηση. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης θα πρέπει να δούμε πώς αντιμετωπίζονται και έρχονται σε επαφή από τις υπηρεσίες μας που είναι επιτόπου στις τρίτες χώρες και πώς ενθαρρύνονται οι υπηρεσίες μας να είναι πιο κοντά όσο πιο κοντά γίνεται με τις οργανώσεις που προσπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε λοιπόν. Θεωρούμε ότι είναι πολύ θετικό μέτρο η δημιουργία μιας ισχυρής διευθύνσεως για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, πράγματι ευχαριστώ βέβαια και τον συνάδελφο Ουγγουρεάνου ο οποίος τόνισε ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης πρέπει να αναλαμβάνει και δράση όπου να είναι. Εν πάση περιπτώσει μια ενισχυμένη ελπίζω ε, πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα να βγει από τη νέα αυτή διεύθυνση. Ε, θα εμείνουμε εμείς σε αυτά τα οποία έχουμε πει εμείς, να υπάρχει δηλαδή μια υπηρεσία που να παρακολουθεί από κοντά την τύχη των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να προσπαθήσουμε να οργανώσουμε καλύτερα και να εξορθολογήσουμε τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές για να καταστήσουμε πιο λειτουργικές τις στρατηγικές σε τοπικό επίπεδο για την πράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χαίρομαι που η κυρία Άστον έκανε μία δήλωση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφωνεί να συναντάτε επίσης με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών που προσπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν αυτό είναι εφικτό. Είναι σίγουρο ότι το θέμα αυτό θα προκαλέσει ενδιαφέρον του κοινού, θα πρέπει να υπάρξει διαφήμιση για τις συναντήσεις αυτές και θα πρέπει επίσης να υπάρχει φυσικά και ε, ε, μια διακριτική παρουσίαση των συναντήσεων αυτών όταν τίθεται να αμφισβητήσει η ασφάλεια των προσώπων τα οποία έρχονται σε επαφή μαζί μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να υπάρξει μια ισχυρή, όπως είπα, διεύθυνση για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Υπάρχει και το θέμα της διαφάνειας σχετικά με τους τοπικούς προσπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της στρατηγικής που θα ακολουθήσουμε απέναντί τους. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε το απόγευμα ε, γύρω από το θέμα αυτό. Χαίρομαι γιατί η Μέρι Λόλερ, η οποία είναι μια εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου που προσπίζεται ε, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διευθύντρια της οργάνωσης Frontline θα είναι μαζί μας να μας παρουσιάσει με περιπτώσει, περιπτώσεις τις οποίες θα πρέπει να υπερασπιστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα είναι η πρώτη μας ομιλήτρια και χαίρομαι που προσκαλώ για μια ακόμη φορά τον κύριο Μούντε της ICON Διεθνής Πόλης Ασύλου όπως ενθυμίστε, είχαμε εμείς ε, αναγνωρίσει το δίκτυο αυτό σαν πρότυπο για την προσπάθεια βοήθειας και προστασίας αυτών που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα τοπικά. Και θα θέλαμε περισσότερες πόλεις να υιοθετήσουν το πρότυπο αυτό και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, εξυπηρετήσει καλύτερα αυτές τις προσπάθειες. Θα ακούσουμε επίσης και από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή για το τι είδου ε, βήματα πρόοδου έχουν γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση και ποιο είναι το μέλλον που προδιαγράφεται. Ε, προς στιγμή δεν είναι σαφές πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Υποεπιτροπή θα συνεργαστεί με τα τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εφαρμόζονται τις πολιτικές αποφάσεις στα θέματα που μας αφορούν. Το θέμα αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί όπως είπα ανάμεσα στα θεσμικά όργανα και χρειάζεται κάποιος χρόνος για να κατασταλάξουν λίγο τα πράγματα. Πάντως, για αυτήν τη συνάντηση θα ακούσουμε και από την κυρία Αρνού, η οποία είναι η νέα διευθύντρια ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πρόθεση της δημοκρατίας. Θα ήθελα οι προσκεκλημένοι μας να μην ξεπεράσουν τα 10 λεπτά στις παρουσιάσεις τις οποίες θα κάνουν Έχουμε καθυστερήσει ε, εκτάκτως κάποιες συζητήσεις. Ξεκινάει η κυρία Λόλερ από την οργάνωση Frontline, πρώτη γραμμή. Ευχαριστώ που μας δίνετε πάλι την ευκαιρία να απευθύνουμε το λόγο στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ένα χρόνο μετά από μια παρόμοια κρόαση και λίγους μήνες μετά την έγκριση από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενός σημαντικού ψηφίσματος για την ευρωπαϊκή πολιτική για την υποστήριξη των υποστηρικτήων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το 2010 σημειώθηκε ε, πρόοδος για την εφαρμογή των πολιτικών για την υποστήριξη των ε, ε, υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων από την Ισπανική και την Βελγική Προεδρία. Η Frontline χαίρεται για, την, για τον διορισμό του αξιωματούχου συνδέσμου για τις επαφές με, τους, με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλιστα και ε, αρμοδίων σε πάνω από 70 χώρες, εκπροσώπων δηλαδή της Ένωσης, που θα επιτρέψει να αναλαμβάνει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία δικαιωμάτων των ε, ανθρώπων που διώκονται. Ορισμένες τώρα έξτρα συστάσεις, έχοντας υπόψη και τις όσες περιλαμβάνονται στις ε, εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για τα εξής θέματα. Πρώτο, η υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων που είναι σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής ανθρώπινων δικαιωμάτων. Την ίδια στιγμή που επανεξετάζει τις πολιτικές της ανθρώπινων δικαιωμάτων που σημειώνονται και μεγαλύτερες δυσκολίες να εξασφαλίσει υποστήριξη με διμερείς σχέσεις τη ατζέντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και όπου η γενική προσέγγιση σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων φαίνεται ορισμένε φορέ να είναι πατερναλιστική και πάντω κατακαιρματισμένη, θεωρούμε ότι με τι νέε αυτέ κινήσει η πολιτική αυτή θα είναι πιο επιτυχημένη μόνο εάν θεωρηθεί ότι διέρχεται όλες τις ε, ε, πολιτικές ε, προστασίας αυτών των δικαιωμάτων η, η γραμμή αυτή που θα πρέπει να αποτελέσει την βάση για τις δράσεις μας. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παγκόσμιο χαρακτήρα. Όπως γνωρίζουμε το λέει και το πρώτο άρθρο της διακήρυξης που λέει ότι όλα τα ανθρώπινα όντα γεννώνται ίσα σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη τους δικαιώματα. Σε ολόκληρο τον κόσμο, λοιπόν, οι υπερασπιστέ των ανθρώπινων δικαιωμάτων αγωνίζονται για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των κοινοτήτων του, διακινδυνεύοντα και την ίδια του τη ζωή. Ο αγώνα του είναι και δικό μα. Η προστασία του, η υποστήριξή του δεν έχει καμία σχέση με την δίθεν δυτική ατζέντα προστασία ανθρώπινων δικαιωμάτων. ή καθήκον τη Ευρωπαϊκή Ένωση να του προστατεύσει και να ε, ανταποκριθεί στι ανάγκε του θα πρέπει να βάλει την προστασία των υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο επίκεντρο των προσπαθειών της. Μόνο τότε θα γίνει πραγματικό μέτρο της εξωτερικής μας πολιτικής, όπως είπε και είπα και εκπρόσωπος ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Δεύτερη σύσταση. Να παρακολουθούνται οι επιμέρους υποθέσεις υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μακροπρόθεσμο, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και να γίνεται προσπάθεια ε, να επιτυγχάνονται πρόοδοι επιτόπου. Έχετε σχετικές ε, υποθέσεις στα έγγραφά σας, όπως Άσκαρα, που συνελήφθη στο Αζερβαϊτζάν και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθεξη και εν, αν και ο ίδιος ο Ομπούτσμαν είπε ότι είναι ε, σαφής παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλο πρόσωπο στην Τεχεράνη. Στην ίδια περίπτωση και σήμερα ακούσαμε ότι άλλο πρόσωπο καταδικάστηκε σε 11 χρόνια κάθεξη και για 20 χρόνια στερείται την ε, δυνατότητα να ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα. Για να εφαρμοστεί τώρα μια τέτοια στρατηγική η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να κάνει σωστό συντονισμό και επιτόπου αλλά και στο κεντρικό επίπεδο για να ξεπεραστούν οι δισταγμοί που εξακολουθούν να βλέπει η Frontline αλλά και άλλες οργανώσεις από πλευρά ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει επίπεδο στο υψηλότερο επίπεδο λέγοντας ως πρόφαση περισσότερο ότι υπάρχουν, γίνεται διάλογο σε υψηλό επίπεδο και ότι δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι. Τώρα ερχόμαστε στην Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων Επιτόπου. Τρίτη σύστασή μου. Ο διορισμός ειδικών αξιωματούχων επιτόπου ανοίγει πολλές δυνατότητες αρκεί αυτοί να έχουν την υποστήριξη των ε, ε, προϊσταμένων τους στις υπηρεσίες τους. Να έχουν τη δυνατότητα να αποκαθιστούν και να διατηρούν επαφές με ε, τις αρμόδιες τοπικές οργανώσεις και να υπάρχουν και βεβαίως αντικαταστάτες τους σε περίπτωση απουσίας τους. Να γίνονται και κατέτος συναντήσεις αλλά καλά προετοιμασμένες μεταξύ των αξιωματούχων αυτών και των οργανώσεων υποστήριξης των ανθρώπινων δικαιωμάτων επιτόπου. Τώρα, για το κεντρικό επίπεδο, χωρίς να συζητήσω τώρα την όλη αρχιτεκτονική δομή της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων, έχω ορισμένε συστάσεις για τον τρόπο που θα πρέπει να λειτουργήσει για το θέμα αυτό. Πέμπτη λοιπόν σύστασή μου. Ε, τα θεμελιώδη θέματα θα πρέπει να γίνονται, να λαμβάνονται υπόψη στο επίπεδο τη εξωτερική ε, υπηρεσία δάσων και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βελτιωθεί ο εσωτερικό ε, συντονισμό και να περάσει μέσα από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Να εξετάζονται λοιπόν οι υποθέσεις, να εξασφαλίζεται μια συνέχεια και ταυτόχρονα και η μελλοντική παρακολούθηση. Και αυτά όλα σε συνδυασμό και με τις προσπάθειες των ειδικών αξιωματούχων. Τώρα, η σύσταση υπαριθμών 6 θα είναι καλύτερη παρακολούθηση εφόσον ειδικό αξιωματούχο διοριστεί για να παρακολουθεί. Η Frontline θεωρεί ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται αυτομάτως στην εντολή και των ειδικών εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνουν δράση, δηλαδή να προσφέρουν feedback και ούτε καθεξής. Έχω και ορισμένες ακόμα ιδέες που μπορώ να σας πω. 7η σύσταση, ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να ενισχυθεί, να γίνει υπόλογο η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων απέναντί του, οι ευρωβουλευτέ να μπορούν να συμμετέχουν σε στοχευμένε δράσει, όπω και στι προηγούμενε περιπτώσει που ανέφερα, και αυτή η προσέγγιση να περάσει μέσα από όλε τι ε, αντιπροσωπείε για ε, σχέσει με άλλα κοινοβούλια, καθώ και όλε τι επιτροπέ του Κοινοβουλίου. Δέκατη σύσταση. Τον Δεκέμβριο είπε η κυρία Άστον ότι συναντήθηκε και θα συνεχίσει να συναντάτε με εκπροσώπους οργανώσεων υποστήριξης ανθρώπινων δικαιωμάτων και ότι αναμένει και από τους συναδέλφους της να πράττουν το ίδιο. Επίσης, οι ανώτατοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συναντώνται συστηματικά με τους εκπροσώπους των ε, οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επισκέπτονται τις Βρυξέλλες. Ένα τη σύσταση. Η Frontline έχει θέσει πάνω από 100 υποθέσεις, ε, διακόπτη κ. Χάουταλα. Διακόπτει η αλλά δεν διακόπτει η ομιλήτρια η οποία μιλεί με ταχύτητα του φωτό. Αν μπορείτε παρακαλώ να μιλήσετε λίγο πιο, να διαβάσετε μάλλον λίγο πιο αργά. Είχαμε λοιπόν θετικές αντιδράσεις σε περίπου 30% ε, των 100 ε, αυτών υποθέσεων που δεν είναι επαρκέ. Θα πρέπει να δίνεται υποστήριξη στου υπερασπιστέ των ανθρώπινων δικαιωμάτων και στι εκκλήσει του για ανάληψη δράσης. Δέκατη σύσταση η Ευρωπαϊκή Ένωση να φτιάξει ένα κώδικα διοντολογία, best practice, που να διαβιβαστεί στις επιτόπου αντιπροσωπείες τη ώστε αυτέ να δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε ορισμένε υποθέσει και στην ασφάλεια των υποστηρικτών των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 11 να γίνονται οι σχετικές παρεμβάσεις στις τοπικές γλώσσες. Δωδέκατη σύσταση, προξενικές θεωρήσεις υπέρ των υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συντάξει ένα εγχειρίδιο για την ε, επεξεργασία των αιτήσεων θεωρήσεων ώστε να διευκολυνθεί η χορήγησή τους σε υπερασπιστές ανθρώπινων δικαιωμάτων και ταυτόχρονα, εν, ε, ε, εν, εν το μεταξύ αυτό, να δοθούν σχετικές οδηγίες στις ε, επιτόπου αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί πρέπει ε, να ε, διευκολυνθεί η χορήγηση προξενικών θυσιορήσεων στους υπερασπιστές ανθρώπινων δικαιωμάτων και η 13η σύσταση θα πρέπει να δοθεί αυτή η δυνατότητα προστασίας και καταφυγίου στους υπερασπιστές ανθρώπινων δικαιωμάτων ήδη από το 2011 και με σχετικές συναντήσεις. Επαναλαμβάνω ότι αυτά θα πρέπει να γίνουν και θυμίζω τον δόκτωρα Μοχάμαντ Άλλη που λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους στο Σουδάν χωρίς ούτε καν προσχηματικά να γίνει δίκη. Είναι η τέταρτη φορά που φυλακίζεται το πρόσωπο αυτό, το πρόσωπο αυτό ο, το οποίο είπε δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αν θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια στην ίδια μας τη χώρα, πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τον κόσμο, με τον λαό, να αγωνιζόμαστε υπέρ αυτού. Χρειαζόμαστε την ενίσχυση της διεθνούς κοινότητας. Χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι μας υπαστηρίζουν κάποιοι άνθρωποι, έστω και αν είναι ηθικά και μόνο. Έχει μεγάλη σημασία αυτή για την ηθική μας ενίσχυση. δεν είναι ορατά τα πρόσωπα αυτά, αλλά νιώθετε να σας κρατούν το χέρι. Αυτά είπε ο ίδιο πριν να φυλακιστεί σα. Πρόεδρο, Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας διαβάσατε. Ε, θα ήθελα απλώ να σας αναφέρω ότι, κατά τη γνώμη μου, πραγματικά ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτό το οποίο προτείνατε. Και έτσι να μπορέσουμε να δούμε ποια είναι η άριστη πρακτική και να γίνει έτσι υποχρεωτικό όλοι να εξετάσουν ότι γίνεται. Τώρα η κυρία Ούλτε. Ο κύριος, συγγνώμη Ούλτε. Έλα τώρα το λόγο για το επόμενο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτέ, αγαπητοί φίλοι, σε ευχαριστούμε που την ευκαιρία να λάβουμε μέρο αυτήν τόσο, σε αυτήν τόσο σημαντική ακρόαση εδώ και 15 χρόνια υποστηρίζουμε όσους δίνουν μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επίσης θα πρέπει να δούμε πώς έχουν σήμερα τα πράγματα γιατί υπάρχουν κάποιες προκλήσεις και έχουμε κάνει κάποια βήματα προς τα εμπρός ώστε να προστατεύσουμε αυτούς ακριβώς τους αγωνιστές για ανθρώπινα δικαιώματα και επίσης θα πρέπει να ε, δούμε κάποια ερωτήματα τα οποία υπάρχουν τόσο ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε για την εφαρμογή ενός νέου συστήματος για αυτές τις ασφαλείς πόλεις για τους ε, ε, αγωνιστές για ανθρώπινα δικαιώματα. Πρώτα πρώτα. Αυτές οι ασφαλείς πόλεις πλαίσια. Το ξεκίνησε αυτό, αυτή η προσθέτει του Ευρωκοινοβούλου το 1995. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, ναι, έκανε επίση ένα σχετικό ψήφισμα και διάφορες αρχέ αρχές, άλλες τοπικές κλπ. Και, έτσι ε, συμμετέσχουν σε αυτή την προσπάθεια ε, άνθρωποι από όλη την Ευρώπη. Ο Σαλμαν Ρώσντι επίση τότε είχε αναδειχθεί, <clears throat> ήταν μια αφορμή και είχαμε τελικά 20 πόλει οι οποίε μπήκαν σε αυτό το πρόγραμμα για, αυτό, για κάποιο είδου προσωρινό ασφαλέ καταφύγιο για του ε, μαχητές για ανθρώπινα δικαιώματα. Επίση έχουμε το κτίριο IPW το οποίο κατέρευσε το 2004 διότι έτσι είχαμε ε, έλλειψη μετά κάποιου φορέα που θα συντονίζει τι σχετικέ ε, ε, τις σχετικές πρωτοβουλίες οπότε άρχισε η διερεύνηση του πώς θα γίνει αυτό και έτσι μπορούμε να δούμε πώς θα υπάρξει ένα δίκτυο αυτό ξεκίνησε και από την 1η 12η του 2005 η ICON, η δική, ο δικό μας φορέας, κινητοποιεί πόλεις, ούτως ώστε να προσκαλούν κάποιους ε, συγγραφείς, κάποιους αγωστήτων με δικαιώματα και επίσης τώρα είμαστε ε, ένας καθιερωμένος οργανισμός εξάρτητος και αυτό ξεκίνησε από την 1η Πρώτου 2010 πέρσι και από την 1η Πρώτου 2011 θα έχουμε πάνω από 30 πόλεις μέλη σε όλη την Ευρώπη και επίσης περιμένουμε την, ε, την Κρακοβία, το Ρεκιαβίκ και την Λιουμπλιάνα, οι οποίοι πρόκειται να μπουν σε αυτή την υπόθεση. Και το Παρίσι επίσης πρόκειται να θεωρηθεί πόλη καταφύγιο για τους διοκόμενους ε, συγγραφείς τώρα για τους αγωνιστές Έχουμε τους ε, bloggers, έχουμε τους ε, δημοσιογράφους, ε, τους συγγραφές, συγγραφείς, ε, ακόμα και σχεδιαστές Mickey Όλοι αυτοί υπάγονται στην κατηγορία των ανθρώπων που θέλουμε να προστατεύσουμε. Μιλάμε για 35 τέτοιους οι οποίοι ήδη βρίσκονται στην, στον καταλογό μας για να προστατευτούν σε κάποια πόλη που εντάσσεται στην ICON. Και έχουμε μια διαδικασία ανάλυση αυτών των αιτήσεων. Ε, έχουμε ένα γραφείο στο Λονδίνο, υπάρχει μια ερευνητική ομάδα και έτσι έχουμε τις συγκεκριμένες προτάσεις για να δούμε ποιοι ανταποκρίνονται στα κριτήρια ε, του καταστατικού της ICON. Ποιοι από αυτούς που έχουν ζητήσει να προστατευτούν. Βασικός στόχος του δικτύου μας είναι να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ του ποιος θα προστατευτεί και σε ποια πόλη. Θα πρέπει να έχουμε γνώσεις και για την πόλη και για τον υποψήφιο. Και για να πετύχουμε θα πρέπει να έχει η πόλη που θα τον φιλοξενήσει ε, τις ε, δυνατότητες να του προσφέρει πράγματα ανάλογα με τις ικανότητες του προστασία και πρόθεση αυτών των ιδεών. Βασικό κριτήριο επιτυχίας και βασικός λόγος γιατί θέλουν να ενταχθούν στην πλατφόρμα πόλεις είναι το ότι θα πρέπει να καταλήξουμε στο να βγαίνει κερδισμένος και ο προστατευόμενος και η πόλη. Έχουμε επομένω συμμετοχή πάρα πολλών δημοτικών και τοπικών αρχών. Βεβαίω και οι προστατευόμενοι αγωνιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, προσφέρουν ε, πολύτιμη εμπειρία, διδάσκουν, συμμετέχουν σε εκδηλώσει, σε προγράμματα ανθρωπίνων δικαιώματα, σε πολιτικέ συζητήσει, γράφουν σε τοπικέ εφημερίδε κλπ. Παράλληλα με αυτέ τι δραστηριότητε, οι φιλοξενούμενοι βεβαίως και ασχολούνται με τους εξόριστους συναδέλφους τους, συναγωνιστές στην χώρα που τους φιλοξενεί και αλλού. Όλα αυτά βοηθούν βεβαίως με την σύγχρονη τεχνολογία και έτσι μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική επικοινωνία και σημαντική επικοινωνία με τα μέσα με πρόσωπα και όλα αυτά μπορεί να γίνουν από όπου κανείς μένει, κατοικεί, όπου βρίσκεται. Πολύ σημαντικό. Κάτι άλλο το πρέπει να δούμε τώρα στα πλαίσια ε, του φόρουμ είναι το εξή. Πώς τα κράτη-μέλη μπορούν να πείσουν κάποιες πόλεις να ενταχθούν σε αυτή την προσπάθεια. Να υπάρξει προετοιμασία, διευκόλυνση της πρωτοβουλίας αυτής και έτσι να έχουμε περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις που θα προσφέρουν καταφύγιο σε αυτά τα πρόσωπα. Παράδειγμα, με, για μια γειτονική μου χώρα. Μέχρι το 2009 δεν είχαμε πόλεις της Δανίας που να είχαν συμμετάσχει σε αυτή την πρωτοβουλία για αγωνιστές δομή δικαιωμάτων και συγγραφείς. Κάποια στιγμή υπήρξε διαφήμιση αυτής της πλατφόρμας και κάποια στιγμή ξεκίνησαν οι σχετικές διαπραγματεύσεις. Το ΔΕ, κοινοβούλιο μας, Ε, απεφάνθη ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί το δικαίωμα για να καλυφθούν αυτά τα οποία ζητεί η ICON. Και τώρα υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο. Και η Δανέζικη κυβέρνηση επίσης συμφώνησε να προστατεύσει και να υποστηρίξει οικονομικά τις πόλεις του δικτύου μας. Η πέμπτη πόλη η οποία προσυπέγραψε συμφωνία είναι η Κοπεχάγη μόλις πριν από ένα μήνα. Και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία επιλογής για την Κοπεχάγη. Εμείς περιμένουμε πώς και πώς να συνεργαστούμε με την Επιτροπή σας, κύριε Πρόεδρε. Και όλους τους άλλους συναρμόδιους. Για το πώς θα υλοποιηθεί αυτή η ιδέα των ασφαλών πόλεων για τους αγωνιστές των δικαιωμάτων. Τώρα θα πρέπει πριν κλείσω να σας πω κάποια άλλα θέματα για να συζητηθούν περαιτέρω όσον αφορά αυτή τη διαδικασία της υλοποίησης της ιδέας μας. Πρώτον, σε ποιο βαθμό θα πρέπει να υπάρχει μια οργανωτική δομή σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κατά πόσο η Άγκον θα μπορέσει αυτές τις προστατευόμενες πόλεις να τις εξυπηρετήσει. Δεύτερο ερώτημα. θα έχουμε ανάγκη ενό πιο συγκεκριμένου οργανισμού, ορισμού για το τι θα πει ε, αγωνιζόμενο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επίση ποια θα είναι τα κριτήρια της επιλογής που θα απαιτούνται σχετικά. Και να δούμε ποιο θα κάνει την επιλογή και ποιο θα αποφασίζει το πόσο αγωνιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πάει σε συγκεκριμένη πόλη. Άλλο ερώτημα. Πόσο κρατά αυτή η προστασία να έχουμε βραχυπρόθεσμη εγκατάσταση ή όχι. Επενθυμίζω ότι για μας ο κανόνας είναι ένα-δύο χρόνια. Μεγάλη πρόκληση. Το τι θα γίνει μετά μια συγκεκριμένη περίοδο, όταν ολοκληρωθεί η περίοδος προστασίας. Άλλο ερώτημα. Τι θα γίνει με το ζήτημα των θεωρήσεων διαβατηρίων. Πώς θα μπορέσουμε επίσης να διευκολύνουμε την παροχή βίζας και να επιταχύνουμε τη διαδικασία χορήγησής της σε κάποιον από αυτά τα πρόσωπα. Κάτι άλλο τώρα. Τι θα γίνει με την ύπατη αρμοστία. Πώς θα μπορέσει να προστατεύσει τέτοιες πρωτοβουλίες Πώς θα μπορούσαμε να έχουμε συντονισμό για να καταλήξουμε σε επαρκή χρηματοδότηση του συστήματος των πόλεων καταφυγίων. Η πόλη μας θα συνεργαστεί με την πόλη των Βρυξελών για το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Παρακαλώ να παρακολουθείτε τι εξελίξει και να έρχεται σε επαφή με του εκπροσώπου τη κάθε φορά που υπάρξει κάποια εκδήλωση εδώ στι Βρυξέλλε ε, θα γίνει αυτό, 24 και 27 Μαρτίου του 2011. Καλώ ορίσατε στην πρωτοβουλία μας. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Θα πρέπει να από τους 8 ή 9 υποψηφίους για την ε, Λευκορωσία ήταν προστατευόμενος σε κάποια πόλη στη φιλανδια 2000-2004 Είχα δε την τιμή να τον δω. Είχε συμμετάσχει πάρα πολύ ενεργητικά στις πολιτικές ζημώσεις των εκλογών του. Και η κόρη του τώρα εκπροσωπεί τις οικογένειες των κρατουμένων. Μεγάλωσε και μένει στην Φιλανδία και έχει ακολουθήσει καλλιτεχνική καριέρα. Επομένως το σύστημα δουλεύει καλά. Τώρα με μεγάλη μου χαρά θέλω να στραφώ στην Βερόνη Καρνό. Να την συγχαρώ για την ανάληψη των καθηκόντων που έγινε λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Θα είναι η διευθύντρια τη νέα διεύθυνση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με μεγάλη μου χαρά. Άκουσα. Και τώρα θα συνεχίσουμε τις επαφές μας σε βάση μηδενική, γιατί αναφέρεται όλο το σύστημα. Ακούσατε τις παρατηρήσεις, τις επικρίσεις για τους ε, αγωνιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πεςτε μας δύο λόγια. Τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά το να έχουμε ένα πραγματικό εργαλείο δημοκρατισμό και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια. Δεν ξέρω αν όλοι χάρηκαν ε, τις δικαιωτικέ εξελίξει. Εγώ πάντω πέρασα πολύ καλέ διακοπέ και για πρώτη φορά εγώ έρχομαι εδώ σαν επίσημη γλώσσα τη υπηρεσία μου γιατί κάτι το νομίζω το οποίο είναι το συμβολικό για την εκδήλωση στο Κοινοβούλιο Έχουμε ξέρετε αυτές τις δύο μονάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα επί τη βάση του των δύο παλαιότερων μονάδων και τώρα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί βεβαίω και υπάρχει αυτή η ιεραρχική δομή ε, και η ιεραρχία ξέρει πώς έχουν αυτά τα προβλήματα Κύριε Χάουταλα, ευχαριστώ και εσά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικότερα για το πόσο σημαντικό θεωρήσατε το θέμα των ε, αγωστόθρωπων δικαιωμάτων, αλλά αυτό και από πλευρά ε, τρομοποιημένων δικαιωμάτων και επίση στο. Ε, πάντοτε δίνετε το παράδειγμα προ μίμηση. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η πολιτική, διότι έτσι μπορούμε να καλύψουμε πραγματικά ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι κάναμε κάποια βήματα προς τα μπρος για την υλοποίηση αυτών των προτάσεων. Και έτσι η αντιπροσωπεία βοηθά να υπάρχει κάποια εκστρατεία επιτόπου. Έχουμε τουλάχιστον μια συνάντηση ετησίως με τους ε, ε, ακτιβιστές των δικαιωμάτων. Έχουμε και τους ε, υπαλλήλους αξιωματούχους συνδέσμους και αυτοί φροντίζουν για τα θέματα συντονισμού. Σε σχέση τώρα με πέρσι, νομίζω ότι καταβάλαμε σημαντικές προσπάθειες. Και τώρα έχουμε 74 όπου είναι δηλαδή πάνω από τις μισές αντιπροσωπείες που ε, έχουν εκπονήσει τέτοιες τοπικές στρατηγικές. Έχουμε ακόμα περισσότερους τέτοιους ανωτέρους υπαλλήλους ε, ε, συνδέσμους, πάνω από 80, οι περισσότεροι είναι στις ε, αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Ε, υπήρχαν λήψεις εκεί, υπήρχαν θέματα ποιότητας στο οποίο στρατηγική και έχουμε ακόμα 62 θέσει τέτοιων συμμετούχων που θα πρέπει να καλυφθούν. Και είπαμε ότι θα πρέπει το τέλο Φεβρουαρίου να έχει ολοκληρωθεί αυτή η στρατηγική, να έχει εκπονηθεί ό,τι χρειάζεται να έχουμε πληρωθεί αυτέ τι θέσει ή να έχει εξηγηθεί γιατί δεν μπορεί να γίνει. Και έχουμε αυτά τα σημεία εστίαση προσπαθειών μα, όπω λέγονται focal points. Είναι αυτά που μα είπατε εσεί στην ομιλία σα. Θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία από τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται συνεργασία και για τις θεωρίες διαβατηρίων, για την υποδοχή, για όλα. Πρόκειται για τις διπλωματικές υπηρεσίες της Ένωσης που ασχολείται. Επίσης έχουμε ε, την αρμοστία που υποστηρίζεται οικονομικά, φτάνει μέχρι το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ και ε, φέτος πάλι πρόκειται αυτή, η, αυτό το ποσό να δοθεί σε κάποιους φορείς και κάποιες οργανώσεις που κάθε μέρα αντιμετωπίζουν δραματικές καταστάσεις. Πάντως για μας είναι θαρρυντικό το ότι στην καινούργια πολιτική για την περιοδο 2011-2013 δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα τα κρατημέλια όσον αφορά τις προτεραιότητες και την προοικοδότηση κατά προτεραιότητα. Ήδη είχαμε κάποιες προτάσεις που ελήφθησαν υπόψη για να καλύψουμε ό,τι ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τώρα, στην επόμενο διαγωνισμό, θα εμπλέξουμε διάφορους διεθνείς φορείς που θα δουλέψουν με τις τοπικές αρχές στενότερα και αυτό το οποίο κάναμε και οι συνάδελφοι την εύκολο να πούνε περισσότερο ότι κάτσαμε και αξιολογήσαμε το πώς γίνεται η, εξε, η εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων. Έχω όλα τα στοιχεία για όποιον θέλει. Συνα, επίσης συνεργασία με την υπατιαρμοστία για τους πρόσφυγες. Στη βάση γραπτών κειμένων προχωρούμε και ήταν πάρα πολύ σημαντικό το να έχουμε συστηματικές επαφές με κυρία Άστον και πολλούς αρμόδιους που Τώρα τα θέματα έχουν όλα ξεκαθαριστεί, που είναι σημαντικό. Και να συνεχιστεί ο συντονισμός με τους διεθνείς φορές, φορείς και υπάρχει επομένως με τον ΟΗΕ, κυρία Σικάκια, είναι η αρμόδια του ΟΗΕ, έγινε συνάντηση Ευρώπης ΟΗΕ και υπάρχει κάτι, κάτι το οποίο το παρατηρήσατε κυρία Πρόεδρε στα πλαίσια έκθεση του Κοινοβουλίου, Είναι δηλαδή το θέμα της ορατότητας. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει από τις αντιπροσωπείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάποιες πολιτικές προσωπικότητες όπως η κυρία Άστον και άλλοι. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα. Είναι αυτό κάτι το οποίο το τόνισε η Μέρη, καθεντήρες γραμμές όσον αφορά αυτούς τους ε, αγωνιστές ανθρώπινα δικαιώματα που δεν είναι γνωστοί. Γιατί δεν έχει γίνει αρκετή δημοσιότητα αυτών των πράσεων. Την αποτελεσματικότητα τώρα έχουμε προοδεύσει, πρέπει να προοδεύσουμε και άλλο και είχαμε αυτές τις άτυπες συναντήσεις μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής και με μη κυβερνικές οργανώσεις θα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε τις τακτές συναντήσεις για να γίνονται ό,τι ρυθμίσεις χρειάζονται. Ακούσαμε και τον τη Σάικον. Θα πρέπει ο ένας να δανειστεί εμπειρίες από τον άλλο για να δούμε πώς θα οργανώσουμε καλύτερα τα πράγματα. να συνδεθούμε και με εσά, να δούμε όλε τι πρωτοβουλίε που έχουν σχέση με τι πόλει καταφύγια. Γιατί έχουμε και κάποιες πρωτοβουλίες που είναι σε επίπεδο μικροοικονομίας και δεν είναι γνωστές. Άρα θα πρέπει να υπάρξει δίκτυο των δικτύων να κάνουμε περισσότερα όσον αφορά κάποιο είδου εσωτερική συνοχή και για τι θεωρήσει. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέχρι σήμερα, όπω ξέρετε, δεν έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε το εγκόλπιο το οποίο αφορά τι θεωρίε διαβατηρίων. Προσπαθούμε όλο ένα περισσότερο να συνεργαστούν τα κράτη-μέλη και τα ξέρουν αυτά οι αντιπροσωπείς. Και νομίζω ότι για τους αγωνιστές με δικαιώματα αυτό θα μας βοηθήσει. Είναι εξωτερική υπηρεσία ακούσαμε τι είπατε. Ακούσαμε τις συστάσεις για τους αγωνιστές των δικαιωμάτων, τους ακτιβιστές. Αυτό που να σας πω είναι ότι βεβαίω, και ακούσαμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά τα σημεία εστίαση τη προσπάθεια. Focal points για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οπότε θα πρέπει και βάσει αυτό να καλυφθούν οι αγωνιστές δικαιωμάτων. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους πολιτικούς συμβούλους της αντιπροσωπείας, οι οποίοι επίσης έχουν και εντολή επικεφαλής της αντιπροσωπείας, οπότε συμβούνταν σε μια κατάσταση υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που ανοίγουν και σε άλλο φορέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι ο φορέας ο πολιτικός και ο φορέας της εργασίας θα συνεργάζονται. Και αυτό πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα για κάποια γενικά θέματα που θα πρέπει από κοινού να τα επιλύσουμε. Πρόκειται για κάποια θέματα τα οποία έχουν τονιστεί στις ε, διαφορετικές συστάσεις. Δεν αφορούν μόνο τους ε, ακτιβιστές δικαιωμάτων, αλλά τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων. Συνεργασία με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και αυτό ανάγεται σε μια γενικότερη προβληματική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και παρόμοια θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την προβληματική για την ελευθερία έκφραση, ελευθερία του τύπου. Πού υπάρχει πρόβλημα σε πολλά κράτη-μέλη. Αυτό φυσικά και αφορά τους ε, ακτιβιστές των δικαιωμάτων. Θα μας προσχωρήσει τα μέσα επόμενα χρόνια. Αυτά θέλω να σας πω. Στη διάθεσή σας. Και όπως προείπα, Χαίρομαι πάρα πολύ για τα νέα μου καθήκοντα, αλλά και ελπίζω θα συνεχίζω να συνεργάζω μαζί σας. Πάντοτε θέλατε έναν ουσιαστικό διάλογο, καλή συνεργασία με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Όποτε υπάρχει διαφωνία, τουλάχιστον γίνεται συζήτηση. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Βερονίκ. Νομίζω ότι η συνεργασία αυτή με τους άμεσα εμπλεκομένους και με τους ε, θεσμικούς παράγοντες θα πρέπει να προωθηθεί. Εφόσον προωθηθεί, θα πετύχουμε ένα νέο επίπεδο στήριξης των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε λίγο χρόνο για συζήτηση και θα δώσω το λόγο στη Μαριτσέ. Ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες εξηγήσεις τις οποίες δώσατε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια στοιχεία των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε έτσι όπως εμφανίζονται σε επίπεδο ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα πολιτικά χαρακτηριστικά αυτών των περιπτώσεων. Στις περιπτώσεις χώρες μέλη, τα Υπουργεία Εξωτερικών είναι υπεύθυνα για τα θέματα αυτά και τα Υπουργεία Εσωτερικών για τις χορηγήσεις θεωρήσεων. Πολλές φορές ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα Υπουργεία Εξωτερικών και Εσωτερικών δημιουργεί προβλήματα. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης βλέπουμε την άνοδο ε, αντιπροσφυγικών αισθημάτων και ακροδεξιών τάσεων και το θέμα της χορήγησης θεωρήσεων είναι ιδιαίτερος ευαίσθητο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους αποσύζευξης αυτών των δύο θεμάτων γιατί αλλιώς φοβάμαι θα οδηγηθούμε αναπόφευκτα σε περιοριστικές και κατασταλτικές πολιτικές, τις οποίες πάνω κάτω δυστυχώς και σήμερα εμπολείς έχουμε. Θα πρέπει επίσης να είμαστε προσεκτικοί, να μην προσπαθούμε να πείσουμε αυτούς οι οποίοι συμφωνούν μαζί μας. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες απόψεις και θα πρέπει τους άλλους να πείσουμε θα πρέπει να λειτουργήσουμε δηλαδή ε, θα έλεγα σε επίπεδο διάδοσης των ιδεών αυτών σε, στα πολιτικά μας κόμματα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το προσπάθησα αυτό. Θέσαμε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις στη Βουλή της Ολλανδίας όπως επίσης και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλεως της Χάγης. Αλλά ο, <clears throat> ο Δήμαρχος της Χάγης διαφώνησε με συνεπώς αν υπάρξει κάποιος τρόπος, αν υπάρχει μάλλον κάποιος τρόπος έτσι ώστε ε, ε, τα, ε, τα, οι δημοτικές και τοπικές αρχές να είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωμένες να ακολουθήσουν τις απόψεις της κεντρικής εξουσίας. Θα πρέπει επίσης <clears throat> να, να τεθεί το θέμα της επεξήγησης των νομικών ρυθμίσεων στις υπηρεσίες που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, των νομικών διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν. Και αυτός θα είναι ένας τρόπος έτσι ώστε να μείνουμε στις ορθές πρακτικές και στα σωστά παραδείγματα. Είχα και άλλη μία ερώτηση προς τους εκπροσώπους των, του δικτύου των πόλεων για το άσυλο. Ποια είναι η διαφορά της δικής τους οργάνωσης με την οργάνωση Shelter Cities, πόλης καταφύγια και τι γίνεται με τις μικρές πόλεις οι οποίες λέγονται πόλεις καταφύγια αλλά από την άλλη είναι τόσο μικρές οι πόλεις αυτές που κάπου αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα αυτά στοχοποιούνται αδίκως. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που έχω να θέσω. Ευχαριστώ. Είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξουν απαντήσεις από τους προσκεκλημένους μας, λέει η Πρόεδρος. Έρχομαι τώρα στον κύριο Πρέντα και μετά στον κύριο Πρόντι. Ο κύριος Πρέντα πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λόουλερ και τον κύριο Λούντε για τις παρουσιάσεις τους. Θα ήθελα επίσης να θέσω ένα ερώτημα προς την κυρία Αρνό. Και εγώ θα ήθελα φυσικά να τη συγχαρώ για το διορισμό της σε αυτήν τη νέα σημαντική θέση. Το κάνατε ήδη κι εσείς. Θα ήθελα όμως, λέγει ο κύριος Πρέντα, να μάθω τι γίνεται με τον διορισμό των υπευθύνων υπαλλήλων συνδέσμων και με τις τοπικές στρατηγικές που ακολουθούνται. Ε, Κυρία Αρνό, γιατί δεν έχουμε ακόμα πετύχει τους στόχους τους οποίους είχαμε, δηλαδή να ολοκληρώσουμε τις στρατηγικές μας σε τοπικό επίπεδο. Γιατί δεν υπάρχουν σήμερα ολοκληρωμένες τοπικές στρατηγικές σε όλες τις περιπτώσεις και γιατί δεν έχουμε παντού υπαλλήλους συνδέσμους ως, ε, ε, όπως θα έπρεπε. Μετά από την απόφαση του Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 για την κυκλοφορία αυτών των καταλόγων των τοπικών στρατηγικών, διαρωτώ με αν θα υπάρξει μια αντίστοιχη συνέχεια και το 2011. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι τέθηκαν αρκετές ερωτήσεις. Οι τελευταίες ερωτήσεις αφορούσαν την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Το λόγο έχει ο κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συζήτηση αυτή που οργανώσατε, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και είναι πολλά τα θέματα που θα ήθελα να θέσω, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την λειτουργία πλέον της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να υπογραμμίσω τις προσδοκίες τις οποίες καλείται να εξυπηρετήσει και προκαλεί η συγκεκριμένη αυτή υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Είναι μια υπηρεσία αναφοράς θα έλεγα και είναι και ένα σημείο σωστής οργάνωσης των δραστηριοτήτων τις οποίες εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε επανειλημμένα αναλάβει στο παρελθόν. Έρχομαι στα θέματα που είχε συμπεριλάβει στην έκθεσή της εδώ η κυρία Χάουταλα, η πρόεδρος. Και να τονίσω ότι υπάρχει και μία προσπάθεια εντατικοποίησης των προσπαθειών μας για καλύτερο συντονισμό των κοινοτικών παρεμβάσεων. πρέπει, οφείλουμε θα έλεγα, να εκμεταλλευτούμε όλα τα δίκτυα τα οποία μας θέτει στη διάθεσή μας ε, η πολιτική δραστηριότητα και αυτά τα περιλαμβάνει έτσι και αλλιώς η έκθεση της Προέδρου μας και να καταστήσουμε πιο αυστηρή την εφαρμογή των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις πολιτικές συμβάσεις και τις εταιρικές συμφωνίες με τρίτες χώρες να υπενθυμίσω επίσης μια περαιτέρω πλευρά η οποία δεν θα πρέπει να αγνοηθεί και η οποία συνδέεται με τις επιπτώσεις των κλιματολογικών αλλαγών τα επόμενα χρόνια στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είχα στο παρελθόν επανειλημμένα να αναφερθώ στο φαινόμενο του climate refugee, του πρόσφυγα για κλιματολογικούς λόγους Μιλάμε για ένα είδος πρόσφυγα το οποίο στο μέλλον θα πολλαπλασιαστεί και προς αυτό τον πρόσφυγα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να σεβαστούμε τα δικαιώματά του και σε επίπεδο διεθνούς δικαίου. Και εδώ τίθεται λοιπόν το θέμα της δυναμικότητας την οποία θα επιδείξουν οι προσπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έτσι ώστε να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων που ασχολούνται με τα θέματα αυτά και οι οποίοι στο μέλλον θα εγκαταλείψουν τις αιστείες τους λόγω ακριβώς των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών. Να εκφράσω επίσης την επιθυμία μου να, πάρω μέρος σε μια, να πάρουμε μέρος σε μια συντενισμένη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δοθούν σωστές απαντήσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία εκφράζουν ε, το συμφέρον που έχουμε όλοι μας για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας. επανειλημμένα εύχεστε πράγματι στο θέμα των κλιματολογικών αλλαγών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε κάποια φορά εδώ λεπτομερέστερα στα πλαίσια του 2011. Ένα ερώτημα τώρα προς την κυρία Αρνό. Μερικές φορές ε, οι ακτιβιστές στον τομέα του περιβάλλοντος που ασχολούνται με τα θέματα των κλιματολογικών αλλαγών και όχι μόνο, χρειάζονται προστασία. Θεωρείται ότι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, υπό το φως όλων αυτών τα οποία είπατε θα μπορούσαν να αναφερθούν στο θέμα των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων όταν συζητάνε θέματα υποδομών για τρίτες χώρες. Είχα τη συζήτηση αυτή με τον Επίτροπο Τίνκερ για το Τουρκμενιστάν. Παράγει πολύ φυσικό αέριο το Τουρκμενιστάν, υπάρχουν πολλά προβλήματα όμως ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα αυτή και πολλούς, πολλοί από αυτούς που θίγονται είναι ακτιβιστές για το περιβάλλον. Και θα πρέπει και ο Επίτροπος για το Περιβάλλον υπεύθυνο να συμμετέχει στις συζητήσεις αυτές, οι οποίες θα πρέπει να είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή των δημοσίων αρχών σε τέτοιου είδους προγράμματα. Ένας από τους πιο γνωστούς πασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν αναγκάστηκε να διαφύγει στο εξωτερικό γιατί απλά έθετε τα θέματα αυτά. Τελείωσαν οι ομιλίες, θα δώσω τον λόγο πάλι στους φιλοξενούμενούς μας. Θα αρχίσουμε πάλι με την κυρία Λόουλερ και μετά θα ακολουθήσουν οι δύο άλλοι. να επιστήσω την προσοχή σας. Αναφερθήκατε στα θέματα των δικαιωμάτων των περιβαλλοντικών. Εμείς έχουμε μία υπόθεση, την οργάνωση που ασχολείται με, τα, με τις περιβαλλοντικές αλλαγές και τις περιβαλλοντικές καταστροφές. Το όνομα της οργάνωσης δυστυχώς δεν το ακούσαμε. Διερωτώμε λοιπόν αν βασιζόμενοι στη συγκεκριμένη περιπτωσολογία μπορούμε να ασχοληθούμε και με το θέμα αυτό υποδειγματικά. Το θέμα της χορήγησης θεωρήσεων τώρα είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Εμείς έχουμε ένα διαρθρωμένο σωστά σύστημα στην Ιρλανδία το οποίο δημιουργήθηκε από την Ιρλανδική κυβέρνηση το 2005. Ο συνάδελφος που είχε θέσει το ερώτημα δεν είναι πια εδώ Λειτουργεί το σύστημα αυτό λοιπόν από τότε. Έχουμε 20 προασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που το χρησιμοποίησαν το σύστημα για να έρθουν στην Ιρλανδία. Έμειναν τρει μήνες το πολύ. Ένας μόνο από τους 20 ζήτησε άσυλο και αυτό συνέβη γιατί η απουσία τους καταδικάστηκαν σε εμφυλάκηση και η κατοικία τους δημεύθηκε. Εν πάση περιπτώσει υπήρξε μια κατάσταση η οποία ήταν αδίωτη για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Αυτό το οποίο λοιπόν θα πρέπει να ενθυμούμεθα είναι ότι οι προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θέλουν να φύγουν και να έλθουν σε άλλες χώρες. Θέλουν να οικοδομήσουν την δίκαιη κοινωνία που ονειρεύονται στη δική τους χώρα. Χρειάζεται όμως μερικές φορές να φεύγουν από τη χώρα τους όταν είναι ακραίος ο κίνδυνος ή όταν έχουν εξαντληθεί πλέον. Φέρνουμε κόσμο, τους δίνουμε τη δυνατότητα να ξεκουραστούν για να ξαναφορτώσουν τις μπαταρίες τους. Έχουμε κάποια προβλήματα τον τελευταίο καιρό με το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ιρλανδία, αντίστοιχα με άλλα τέτοια ε, ε, Υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικών σε άλλες χώρες αλλά συμφωνούν με τη μέθοδο που ακολουθούμε σε πιλωτική βάση. Έχουμε ένα καλό πρόγραμμα, χορηγούνται οι βίζες, οι θεωρήσεις γρήγορα και δίδουμε τις εγγυήσει έτσι ώστε να υποστηρίξουμε αυτούς που προσπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο είναι μαζί μας. Σε επίπεδο επιμελητιακό είναι απλή υπόθεση, Βγάζουμε τη θεώρηση, τη βίζα, στέλνουμε επιστολές στην πρεσβεία όπου θα κάνουν την αίτηση, online συνήθως όταν είναι διαθέσιμη η μέθοδος αυτή και όταν έρχεται το συγκεκριμένο πρόσωπο η αστυνομία στο αεροδρόμιο έχει το όνομά του, το διαβατήριό του κτλ. Και τα τελευταία χρόνια εννέα χρόνια ε, που λειτουργεί το Frontline ε, εκδόθηκαν 550 τέτοιες θεωρήσεις και μόνο από 5 από τους 550 ζήτησαν πολιτικό άσυλο. Αυτό δείχνει ότι οι προασπιζόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα θέλουν κυρίως να ζουν στις χώρες τους. Πράγματι αυτά τα οποία ακούσαμε από την Ιρλανδία είναι μια θα έλεγα βέλτιστη πρακτική η οποία είναι προς μίμηση, είτε συμφωνούμε είτε όχι. Είναι κάτι το οποίο σαν πρότυπο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και από τους άλλους. Την προηγούμενη εβδομάδα ε, υπήρξε ένα σημαντικό πρόβλημα με το Υπουργείο Εσωτερικών μιας χώρας που αρνήθηκε να χορηγήσει βίζα σε, δεν θέλω να ονοματίσω ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έδωσαν τις θεωρήσεις που έπρεπε να δώσουν ε, για την εκπαίδευση κάποιων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Λοιπόν, ο κύριος Μούντε είναι ο δεύτερος προσκεκλημένος. Νομίζω ότι δύο ενδιαφέροντα ερωτήματα ακούστηκαν προηγουμένως. Θα απαντήσει στο ένα η συνάδελφός μου, στο δεύτερο. Το πρώτο είχε το εξής περιεχόμενο. Αν υπάρχει δηλαδή διαφορά ανάμεσα στο δίκτυο που εκπροσωπούμε εμείς, το ICON, και το δίκτυο πόλεων καταφυγίων. Πρόκειται για σύμπτωση. Το γεγονός δηλαδή ότι η δική μας οργάνωση είναι νέα Αναπτύσσεται όμως και ταυτόχρονα η πρωτοβουλία των πόρων καταφυγιών επίσης αναπτύσσεται. Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς εμπειριών από την ICON στο Shelter City που είναι η πόλη καταφύγιο. Εμείς αρχίσαμε και συνεχίζουμε να είμαστε ένα δίκτυο πόλεων καταφυγίων με ευρύ ορισμό βέβαια προσώπων που μπορούμε να δεχόμαστε, που μπορεί να είναι δημοσιογράφοι, μεταφραστές, ακόμη και α, α, σκηνοθέτες κινηματογραφικών ταινιών και ούτω καθεξής. Κάθε δηλαδή άνθρωπος, κάθε υπο, υπερασπιστής ανθρώπινων δικαιωμάτων που είναι υποχρεωμένος ή υποχρεωμένη να εγκαταλείψει την χώρα του μπορεί να απευθυνθεί σε εμά και θα αντιμετωπίσει θέματα βέβαια αργά ή γρήγορα στη χώρα του ελευθερίας έκφρασης και αυτό μας οδηγεί σε στενή συνεργασία και στο μέλλον θα πρέπει να κρυφεί. Χρειαζόμαστε μια νέα δομή, ρωτήσατε, ή μπορούμε να βασιστούμε σε αυτές που υπάρχουν. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι γιατί έχουμε δεχτεί προσκλήσεις να, να, να συμμετάσχουμε σε τέτοιε συζητήσεις και θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία με όλους τους άλλους εταίρους για να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του δικτύου αυτού ε, πόλεων καταφυγίων για τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και για το άλλο ερώτημα, η Ελίζα, αν επιτρέπετε, ναι, για μικρότερες πόλεις όπου υποδεχόμαστε κυρίως ε, συγγραφείς και άλλε τέτοιου υπερασπιστές ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα για την ώρα. Όταν κάποιος ζητεί, κάνει αίτηση δηλαδή να τον δεχθούμε σε μια τέτοια πολύ καταφύγιο γνωρίζουμε ότι αυτό είναι η ίστατη καταφυγή του. Γνωρίζουμε ότι έχει ήδη αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Εμείς είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση ονομάτων ή ε, ποια πρόσωπα βρίσκονται ε, στις λίστες αναμονής μας. Όλα αυτά τα χειριζόμαστε ως εμπιστευτικές πληροφορίες. Και κάνουμε πάντοτε μια αξιολόγηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων εάν δημοσιευθεί το όνομα αυτό και ζητούμε από το ίδιο το πρόσωπο να πει εάν θα ήθελε το όνομά του να δημοσιευθεί όταν φτάσει σε μία από τις πόλεις καταφύγια και συχνά τα πρόσωπα αυτά δεν επιθυμούν να δημοσιευθούν τα ονόματά τους. Σε ό,τι αφορά τώρα τις βέλτιστες πρακτικέ σχετικά με τι προξενικέ θεωρήσει, η ιδανική κυβέρνηση πρόθεσε νομοσχέδιο για την ε, χορήγηση προξενικών θεωρήσεων σε περιπτώσεις όπου προσκαλούν οι πρασπιστέ ανθρώπινων δικαιωμάτων κάποιες πόλεις στη Δανία, μικρές πόλεις, ε, που είναι ε, οι προξενικές αυτές θεωρήσεις διάρκεια δύο ετών δίνουν το δικαίωμα να εργαστούν αλλά μόνο, μόνο ως ε, υποστηρικτές ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δηλαδή μέσα σε, ε, στα πλαίσια αυτά. Όχι οποιαδήποτε δουλειά. Δεν μπορούν να ασκήσουν οποιαδήποτε δουλειά ή επάγγελμα, αλλά μόνο ε, να εργαστούν μέσα στα πλαίσια αυτά. Μάλιστα, Χάουταλα, πρόεδρο. Σα ευχαριστώ. Τα σημειώνουμε αυτά που μας είπατε. Η κυρία Αρνό τώρα, Βερονίκ. Σας ευχαριστώ κυρία Χάουταλα. Σχετικά με το θέμα του ορισμού και της ε, ευαισθητοποίησης πρέπει να γίνει ξεκάθαρα διάκριση ανάμεσα στους υπερασπιστές ανθρώπινων δικαιωμάτων και σε αυτούς που ζητούν άσυλο. Πρέπει να γίνει προσπάθεια και μέσω των πολιτικών κομμάτων προς την κατεύθυνση αυτή. Δεύτερο, Υπάρχουν ορισμένε χώρε μέλη που έχουν καλή πρακτική, όπω η Ιρλανδία, όχι όμω μόνο, υπάρχει και η Σουηδία, οι κατοχώρε, η Ισπανία. Πάλι πρέπει να εξετάσουμε ποιον τρόπο αυτέ οι καλέ πρακτικέ μπορούν να αποτελέσουν πηγή εμπνεύσεω και για άλλε χώρε μέλη. Το δεύτερο ερώτημα που τέθηκε ήταν σχετικά με τον ορισμό των υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων και όπως είπαν οι κύριοι Πρόντι και Χάουταλα για τις ε, σχέση με, γιατί, για τις ειδικότερες ενέργειες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει ο ορισμός αυτός να είναι γενικός, αρκετά γενικός και να συμμορφώνεται με τον ορισμό των ΗΕ του 1998. Στην κατηγορία αυτή έχουμε ένα ευρύ φάσμα που καλύπτουμε πολλούς υπρέψεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι ε, πάσχουν ε, πλήττονται από ε, παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, ε, δικαιωμάτων του πολίτη, αλλά και περιβαλλοντικών, έλλειψης ελευθερίας έκφρασης, του, της ελευθερίας του συνέρχεστε ή του συνεταιρίζεστε. Αυτά τα πράγματα λοιπόν θα πρέπει να παραμείνουν σχετικά στα πλαίσια ενός ευρέως ορισμού. και σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα και σε ό,τι αφορά τα πολιτικά δικαιώματα. Η ερώτηση πρέντα, γιατί δηλαδή γιατί όλες οι χώρες όπου υπάρχουν διπλωματικές αντιπροσωπείες για 22 χώρες δηλαδή όπου δεν έχουμε εκπροσώπηση γιατί δεν έχουν όλες αυτές οι χώρες μια στρατηγική. Μα εδώ υπάρχουν τέσσερις λόγοι. Πρώτον, έλλειψη δυναμικού αντιπροσωπιών. Υπάρχουν ορισμένε χώρες Ανατολικό Τιμόρ, για παράδειγμα, όπου έχουμε πάρα πολύ μικρή δυνατότητα εκπροσώπησης. Επίσης, καταπιστικά καθεστώτα το Ιράν, το Σουδάν, η Ερυτρέα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να συναντηθεί κανεί με υπερασπιστέ ανθρώπινων δικαιωμάτων και να αναπτύξει μια στρατηγική. Οι συνάδελφοί μα πάντω προσπαθούν. Το Ιράν όμω είναι μια τέτοια περίπτωση όπου δεν υπάρχει τέτοια ε, ικανότητα εκπροσώπηση. Άλλο πρόβλημα είναι χώρε όπου υπάρχει ανυπαρξία κοινωνίας των πολιτών ή αδυναμία εντοπισμού Κοινωνία των πολιτών, είτε διότι είναι πάρα πολύ καταπιστικά τα καθεστώτα, είτε λόγω ιστορικών λόγων, για παράδειγμα Μαδαγασκάρη. Τέλος, μπορεί να έχουμε και πολιτικές διαφορές μεταξύ χωρών μελών και δυσκολίες σε ό,τι αφορά την εκπόνηση μιας στρατηγική για τη συγκεκριμένη χώρα. Για παράδειγμα, μια χώρα είναι το Μαρόκο. Με το Μαρόκο και ιδίω σχέση με την Δυτική Σαχάρα και έχουμε πρόβλημα και με τη Βραζιλία και με τη θέση της Βραζιλίας ως ε, διεθνούς εταίρου. Έχουμε λοιπόν διάφορες κατηγορίες δυσχεριών. Σε ό,τι αφορά τώρα την δημοσίευση, δύο πράγματα έχω να πω εδώ. Πρέπει να υπάρχει ταυτοποίηση και δημοσίευση των ονομάτων των προσώπων που είναι οι ε, τοπικοί εκπρόσωποι μας. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι μπορούν να είναι οι άμεσοι συνομιλητές των ενδιαφερομένων. Αυτό το έχουμε συζητήσει και με τις χώρες μέλη και βέβαια υπάρχουν και προφανείς λόγοι ασφάλειας καθώς και το γεγονός ότι θέλουμε να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή ευκαμψία στη συνεργασία μας με τις χώρες μέλη, γιατί τα θέματα αυτά είναι και πολύ ευαίσθητα. Σε ό,τι αφορά το τι θα, μπορούσαμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε εν προκειμένου. Δεν έχουμε πρόβλημα να διαβιβάσουμε και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων αλλά και στην κυρία Χάουταλα την λίστα αντιπροσωπιών και εκπροσωπήσεων όπου υπάρχει ένα σημείο εστίασης, ένα focal point, αλλά και μια στρατηγική. Έχοντας υπόψη όμως ότι θα έχουμε τον πλήρη κατάλογο μέχρι τα τέλη του Φεβρουαρίου. Και εν προκειμένου, μάλλον, α, μια στιγμή υπάρχει και κάτι ακόμη. Η ανακοίνωση στο Κοινοβούλιο των ίδιων των στοιχείων στρατηγικής. Γνωρίζω ότι αυτό σας ενδιαφέρει πολύ και με εσά κύριε Χαουταλά πρέπει να συζητήσουμε τη ρύθμιση για τις εμπιστευτικές πληροφορίες. Είναι σημαντικό να έχετε πρόσβαση, αλλά σήμερα δεν είμαι σε θέση να σας υποσχεθώ τίποτε περισσότερο από την διαβίβαση του καταλόγου. Σας ευχαριστώ κυρία Αρνό. Νομίζω ότι απαντήσατε ορθά σε όλες τις ανησυχίες που εκφράσαμε και για την ανάγκη επίσης περαιτέρω συνεργασίας. έχω κι εγώ το εφιάλτη ότι ο Julian Assange μπορεί ε, να ε, αποκτήσει πρόσβαση σε κάποιες από τις εμπιστευτικές πληροφορίες. Ναι, μεν είναι αξιοθαύμαστη η πρωτοβουλία που έχει αναλάβει με την Wikileaks, αλλά θα πρέπει να κατανοεί πλήρως την κατάσταση των προσώπων αυτών που των προσώπων αυτών που δεν ε, θα πρέπει να βγουν στο φως της δημοσιότητας. Νομίζω ότι ε, εδώ μπορεί να λήξει η συζήτηση αυτού του σημαντικού θέματος οροσίμου στις σχέσεις μας με τα άλλα θεσμικά οργανά αλλά και με την ε, κοινωνία των πολιτών για να βρούμε τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας με τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων και είμαι βεβαία ότι και οι συνάδελφοί μου της Γραμματείας της Επιτροπής μας έχουν σημειώσει προσεκτικά τις γνώμες που εκφράστηκαν και θα εξετάσουμε τα εναπομένοντα θέματα με λεπτομέρεια. Θα ζητήσουμε και από την Γραμματεία να οργανώσει την συνέχεια της σημερινής συνεδρίασης. Ελπίζω λοιπόν θα μπορέσουμε να παραμείνουμε σε επαφή μαζί σας και να συνεχίσουμε την αγαστή συνεργασία μας. Χρειάζεται και αυτό το όργανο διαθεσμικής συνεργασίας που να αντιμετωπίσει το θέμα υπό τις πολλές πτυχές του. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλες και όλους πολύ και για την εξαιρετική ε, συνεργασία σας στην ε, εκπόνηση της ε, συνεργασίας αυτής. Τώρα, ας έρθουμε να συζητήσουμε το τι γίνεται με τη λειτουργία της υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Έχουμε τον Τιτ από το δίκτυο για την δημοκρατία. Ήδη είναι θέμα σημαντικό το οποίο το έχουμε ε, φίξει για να δούμε τι γίνεται όσον αφορά το οργανόγραμμα της υπηρεσίας αυτής και θα πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει να υπάρξει συμμετοχή από την κοινωνία των πολιτών και αν δεν υπήρχε δεν είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Ο Ντέιβ Νίκος όμως να λάβει το λόγο για να μας πει δύο λόγο όσον αφορά το τι πρεσβεύει αυτό το δίκτυο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας και, και η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν κάποιες σχετικές φήμες σε σχέση με το τι γίνεται όσον αφορά αυτή την εξωτερική υπηρεσία, την υπηρεσία της δράσης, για το τι δομή θα λάβει. Πάντως θα πρέπει να μας ικανοποιούν τα όσα έχουμε πετύχει, θα πρέπει να μας ικανοποιεί το ποιοι έχουν μέχρι τώρα κληθεί να εργαστούν εκεί. Εδώ, πλευρά Κοινοβουλίου, θα πρέπει να δούμε το ότι είναι δυνατόν να έχουμε αυτή, αυτή την ομάδα εργασία του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε και εγώ περιμένω πώ και πώ να ακούσω. Να ακούσω τι γίνεται. Να μας, αυτά που είπε ο κύριος Έγκελμπερτ Τόιρμαν από την Αυστρία. Δεν ξέρω, συμφωνεί με αυτά τα οποία εμεί πρεσβεύουμε, συμφωνεί με του δικού μα στόχου. Για να ακούσουμε τώρα. Πρώτα τον κύριο Νίκολ, με την κυρία Αρνό. Πώ έχει η κατάσταση και ε, πώ λέτε, τι προκλήσει που αναδύονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την ευκαιρία που μα δίνετε στο δίκτυό μα να επανέλθουμε και να σα μιλήσουμε για την υπηρεσία εξωτερική δράση. Όπως είπαμε, ε, έχουμε ένα σωρό άλλους ε, φορείς που ε, όλο ένα και περισσότερο ανησυχούν όσον αφορά το τι θα γίνει ε, στη συνέχεια του 2010, γιατί είπαμε ότι αυτή η υπηρεσία εξωτερική δράση θα αποκτήσει κάποια δομή και τράβηξαν πολύ χρόνο να ληφθούν κάποιε αποφάσει. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου πληροφορίε για του εμπλοκόμενου και επομένω όλο ένα και περισσότερο ανησυχούμε από πέρσι και μετά επίση. Είχαμε κάτσει και τα είχαμε συζητήσει και κρατούσαν αυτές οι συζητήσεις ε, για το πόσο μπορούμε τελικά να, μπορούμε να αναλάβουμε δράσεις σε τέτοιες περιπτώσεις γιατί, ε, γιατί τελικά αφού δεν υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις είναι αρνητικό αυτό για τη δράση μας όλο είναι και χειρότερα όμως να ήρθαν δύο καλά μαντάτα περί τα Χριστούγεννα πρώτα πρώτα τελικά ε, δημοσιεύθηκε το, η τελική εκδοχή του οργανογράμματος όπως είπατε έχει, έχει, έχει μια διεύθυνση για ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία εκεί έχουμε τρία τμήματα και υπάρχει ένας μόνιμος επικεφαλής και τελικά η Κόχομ πρόκειται επισήμως να αναγγείλει πρόγραμμα εργασίας φέτος και ακριβώς για αυτά τα δύο ζητήματα θεωρούμε ότι και εσείς ε, διάφοροι ευρωβουλευτές βοηθούν και βοήθησαν ιδίω κατά τις συζητήσεις στο Στρασβούργο τότε που ήρθε η Βαρόνη λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Αυτό ήταν όλο ένα και πιο, και πιο ε, κρίσιμο γιατί τότε πρέπει να ληφθούν κάποιε αποφάσεις. Τώρα, δεν ξέρω αν σας εκπλήσει το ότι δεν τέλειωσε η υπόθεση. Γιατί αναδύονται τώρα πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα αφού δημοσιεύθηκε το οργανόγραμμα και να σας πω κάποια σημεία και να τα συζητήσουμε μετά. Να, έχουμε πέντε τομείς όπου έχουμε ερωτηματικά πρώτα-πρώτα τις ε, θέσεις υψηλού επίπεδου στην υπηρεσία. Θα θυμάστε ότι ζητούσαμε να υπάρχει ατομική ευθύνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη, στο, στο Συμβούλιο Διαχείρισης, στο Διοικητικό Συμβούλιο τέλο πάντων της υπηρεσίας. Ατομική ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα υπάρχει ατομική ευθύνη για μία θέση. Όμως Ούτε ξέρουν ποιος είναι, ούτε αυτή η υπόσχεση δόθηκε επισήμως και δημοσία. Και δεν μας είπαν καν ποιος θα είναι ο επικεφαλής αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πολυμερή ζητήματα τα οποία θα είναι αρμοδιότητες της εξωτερικής υπηρεσίας. Είναι πολύ σημαντικό όποιος οριστεί εκεί να είναι έμπειρος, να καταλαβαίνει από διεθνέ δίκαιο, γιατί αυτό αφορά το χαρτοφυλακείο του. Μάλλον δεν βρήκανε κάποιον που να έχει τα πρώτα προσόντα και εμπειρία. Οπότε θα πρέπει η διαδικασία αυτή να διευρυνθεί, να κάτσουν να λάβουν υπόψη ποιοι ήδη εργάζονται με αυτά τα προσόντα σε Κομισιόν και Συμβούλιο. Επίσης υπάρχει αυτές τις υψηλές Έχουμε τι εκθέσει αντρικένη και λοιπά. Τα έχουν πει και διάφοροι ευρωβουλευτές. Υπάρχουν ειδικοί απεσταλμένοι εκπρόσωποι για θέματα γυναικών, για διεθνέ δίκαιο, για δικαιώματα ανηλίκων κλπ. κλπ. Δεν ξέρουμε αν θα προβλέπετε κάτι τέτοιο στο μέλλον. Επίσης, όσον αφορά την δομή της υπηρεσίας τη Βρυξέλλες. Από ό,τι κατάλαβα, αυτό το οργανόγραμμα είναι μία μόνο αρχική φάση. Επόμενο εξάμεινο χρόνο, βάσει της κτήθης εμπειρίας, θα χτενιστεί. Και θα έχει την ευκαιρία το Κοινοβούλιο, αλλά και οι μη κυβερνικές οργανώσεις να δουν το πώς δουλεύει στην πράξη αυτή η υπηρεσία. Να διατυπώσουν προτάσεις, πώς μπορεί να βελτιωθεί η λειτουργία της, μια που δεν έχει αποκρισταλωθεί η κατάσταση και να δούμε αυτές, τα, αυτά τα τρία τμήματα της διεύθυνσης πώς θα λειτουργούν. Και αν είναι δυνατόν κάποιοι πάρει από την Κομισιόν εκεί να πάνε να δουλέψουν, ε, τι θα γίνει. Εκεί πέρα υπάρχουν κάποιοι φόβοι. Τι γίνεται με τις ε, Πώ θα υπάρχει συντονισμό τέλο μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών τη αυτή τη υπηρεσία, των τμήματων και πώ θα συντονίζονται, πώ θα λαμβάνουν αποφάσει με κάποια συνέπεια. Είπαμε δεν θα υπάρξει αύξηση προσωπικού, ε, θα πάρουν υπαλλήλου από συμβούλιο και κομισιόν. Θα αναλυθούν δηλαδή κάποιε αρμοδίτες που είχαν οι προεδρίες. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ούτε προσωπικό ούτε πόρου για τον χρόνο. Ήδη είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία κοχόμ στις Βρυξέλλες. Και να έχει έναν σταθερό επικεφαλής πρόεδρο. Όμως τα κράτη-μέλη δεν έχουν πιστεί ακόμα ότι αυτό είναι απαραίτητο. να κάτσουμε εμεί και να αξιολογήσουμε τώρα ποια είναι τα πλεονεκτήματα, ποια θα είναι η προσθεμένη αξία που θα προκύψει. Σε σχέση και με το τι θα γίνουν άλλε πολιτικές της Ένωση Τρίτον, για τι αντιπροσωπείε. Αυτό το οργανόγραμμα αφορά εδώ τη βασική υπηρεσία της Βρυξέλλε και όχι τις αντιπροσωπείε. Άρα, ακόμα δεν ξέρουμε πώ θα εξασφαλιστεί το ότι θα υπάρχει κάποιο ασχολείται με ανθρώπινα δικαιώματα στι αντιπροσωπείε. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απαραίτητη συνεργασία μεταξύ αντιπροσωπιών και πρεσβειών ΕΕ. Έχουμε 100 Έχουμε, έχουμε τόσο κάποιου στι 103 αντιπροσωπείε που ασχολούνται με ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά θα πρέπει παντού να υπάρχει κάποιο που ασχολείται με ανθρώπινα δικαιώματα. Σε όλε τι αντιπροσωπείε και βέβαια να δοθεί προτεραιότητα σε κάποιες χώρες για τέτοιους αξιωματούχους υπαλλήλου. Θα πρέπει βέβαια να δοθεί καλύτερος ορισμός του τι είναι σημείο εστίασης δράσης. Focal point. Είπαμε θα διαδεχθούμε το ρόλο των προεδριών, τι γίνεται με τις πρεσβείες. Να διευκολύνουμε τις πρεσβείες όπου έχουν τις γνώσεις, το προσωπικό, τη δυνατότητα να ενεργήσουν, να τις βοηθήσουν. Η υπηρεσία όπως έχει σήμερα αποτελεί ντροπή για την Ένωση όσον αφορά την ισορροπία υπαλλήλων από τα δύο φύλλα. Δεν λαμβάνει υπόψη τη δέουσα ισότητα των δύο φύλων. Κάναμε πρόκειται στο κοινοβούλιο, αλλά τις απονεύρωσε ή είπε το κοινοβούλιο. Να ληφθεί λοιπόν υπόψη πρότασή μα και όσον αφορά του επικεφαλεί των προσφύγων στο μέλλον. Τέλο, τι ίδια με την αναθεώρηση τη πολιτική για ανθρώπινα δικαιώματα. Πάρα πολύ βασικό το τι έγινε πέρσι. Πέρσι είπαμε ότι θα πρέπει να διαμορφωθούμε, να διαμορφώσουμε κάποιε στρατηγικέ τα είπε αυτά η Βαρονή Άστον στην Ολομέλεια πριν τα Χριστούγεννα. Να δούμε ποιοι θα εμπλακούν, αν, αν κάποιοι τα τρομερά δικαιώματα θα συμμετάσχουν, αν το κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει τη γνώμη του τι θα κάνουν οι άλλες, τι θα κάνουν τα άλλα θεσμικά όργανα, αν το κοινοβούλιο θα ελέγξει τα όργανα, αν η ΚΟΧΟΜ επίσης θα στελεχωθεί από τα άλλα θεσμικά όργανα. Επίσης, ακόμα δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα γίνει η αναθεώρηση της περσινής πολιτικής για ανθρώπινα δικαιώματα, πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η αναθεώρηση, γιατί θα πρέπει να πάμε να συνοηθούμε να βρούμε τη Βαρόνια στον πριν τα Χριστούγεννα γιατί όπως ξέρετε, η τελευταία ανακοίνωση ανθρώπινων δικαιώματα ανάγεται στο 2001. Ε, όμως τώρα είναι απαρχιωμένη, τουλάχιστον όσον αφορά το ότι θα πρέπει όλοι να έχουν κάποιο έγγραφο που να αναφέρεται ποιε είναι οι αρμοδιότητες, ποιε είναι οι ευθύνε, όλα αυτά και να ορίζονται. Να έχουν ξεκαθαριστεί τα πράγματα πολύ περισσότερο από ό,τι γίνεται σήμερα. Το τελικό σημείο αφορά τις προσδοκίες που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσδοκίες οι οποίες απευθύνονται από το δίκτυο προς το Κοινοβούλιο καλύτερα να το πω. Βασική μας προσδοκία είναι να υπάρξει συνέχιση ε, και προσοχή στις αποφάσεις οι οποίες ε, ε, έχουν ληφθεί σύμφωνα με την έκθεση Αντρική Ένε. Μετά από τη δημοσίευση του οργανογράμματος θα υπάρξει περισσότερη περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε εσά Πρόεδρε και στη Βαρόνια Άστον σχετικά με το πόσο θα εφαρμοστούν οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση Αντρική ΕΝΕ. Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως και η ΜΚΟ θα πρέπει να μπορούν να παρακολουθήσουν στενά τον τρόπο λειτουργίας της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης τους επόμενους μήνες και να υπογραμμίσουν τις πιθανές αδυναμίες. Όπως έχω ήδη πει, το 2010 είδαμε να υπάρχει μια χειροτέρευση του τρόπου εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα μέσω της σύγχυσης που δημιουργήθηκε με τις νέες δομές της μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Δεν μπορούμε να σας πούμε εμείς ακριβώς τι έχει συμβεί με την υποστήριξη την οποία αναμέναμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια σε τοπικό επίπεδο. Απλά φέρνουμε το παράδειγμα της Τινησίας όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν απολύτως σιωπηλή σε σχέση με την σημαντική καταστολή των ανθρώπων που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί. Είμαστε απογοητευμένοι γιατί η χειροτέρευση αυτή της ε, δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπογραμμίστηκε στη συζήτηση στην Ολομέλεια πριν από τα Χριστούγεννα. Ένα τυχαίο παρατηρητή αυτή τη συζήτηση. θα θεωρούσε ότι τα πράγματα βαίνουν καλώ όπω και την προηγούμενη περίοδο. Αντίθετα χρειάζεται και οι βουλευτέ χρειάζεται να είναι σε στενή επαφή και να ελέγχουν τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα για να δουν αν εφαρμόζουν διπλά μέτρα και σταθμά. Και τέλος, οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να συνεργάζονται με τους βουλευτές των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Οι βουλευτές των κρατών μελών θα πρέπει να γνωρίζουν ποιες είναι οι νέες δομές και οι νέες ευθύνες και τις συγκεκριμένες νέες υπηρεσίες αλλά θα πρέπει και οι βουλευτές από τα κράτη-μέλη να μπορούν να πιέζουν έτσι ώστε να λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο. Και αναφέρομαι εδώ στις προτάσεις της κυρίας Αντρικίενε. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο λοιπόν Πρόεδρε, να στείλετε μία επιστολή στους Προέδρους των Αρμοδίων Επιτροπών των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών σχετικά με την προώθηση των θέσεων της εκθέσης Αντρικίενε σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριε Νίκολς για την δήλωση την οποία έκανες εξ του δικτύου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Πάρα πολύ συνοπτικά θα ήθελα να πω ότι εμείς έχουμε προκλήσεις και στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προτείνουμε ε, θα έλεγα συντεταγμένες ε, πολιτικές ε, γραμμές για να βοηθήσουμε και τους συναδέλφους ε, που προσπίζονται, που ταξιδεύουν μάλλον με τις αντιπροσωπείες και έρχονται σε επαφή με προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι κάτι το θετικό. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν συνάδελφοι που από μόνοι τους δεν θέτουν τα θέματα αυτά στις επαφές που έχουν σε τρίτες χώρες και δεν είναι διατεθειμένοι να δεχθούν όλους όσους θα πρέπει να συναντήσουν. Σχετικά με τα κοινοβούλια των κρατών μελών, η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά εθνικά κοινοβούλια τα οποία εμπλέκονται άμεσα στις πολιτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς όπως και άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές είχαμε την δυνατότητα να οργανώσουμε κοινέ συναντήσεις με τους συναδέλφους από τα κοινοβούλια των κρατών μελών και μετά από προσεκτικές συζητήσεις που είχαμε για την επερχόμενη αναθεώρηση και για τον τρόπο με τον οποίο τα κοινοβούλια αυτά μπορούν να πιέσουν τα Υπουργεία Εξωτερικών και άλλα Υπουργεία των κυβερνήσεών τους να φέρουν εις πέρα στις ανηλυμένες υποχρεώσεις τους, είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν ακόμα περισσότερο στο μέλλον και όχι να μιλήσουμε μόνο για θέματα, θα έλεγα, περισσότερο θεωρητικά. Σχετικά τώρα με την προτινόμενη αναθεώρηση, τα ήθελα, ελπίζω, ονειρεύομαι ότι αυτή η επερχόμενη αναθεώρηση θα είναι σε βάθος, δεν θα κάνει αποκλεισμού και θα είναι ιδιαίτερος λεπτομερής. Νομίζω ότι ίσως χρειάζεται μια διαφορετικού μορφή, διαφορετικής μορφής επικοινωνία από πλευράς της, ε, ε, του υπάτου εκπροσώπου, που εκπροσωπεί βέβαια και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η ανακοίνωση αυτή θα πρέπει να έχει σαν στόχο και το, Υπουργείο, και το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών. Περιμένω λοιπόν με πολλή επιθυμία τις προοπτικές αυτές στα πλαίσια της νέας διεύθυνσης της οποίας έχει διοριστεί η ηγέτης πλέον η κυρία Αρνό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εσάς προσωπικά και όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλες τις ΜΚΟ οι οποίες ε, έδωσαν ε, μεγάλες μάχες όχι μόνο για να υπάρξει το λεγόμενο mainstreaming σε εισαγωγικά αλλά για να υπάρξει και μια συλλογή συγκεκριμένης ε, εμπειρογνωμοσύνης θα έλεγα τελικά υπήρξε μια ξεκάθαρη πλέον δομή με την οποία θα μπορέσουμε να δουλέψουμε. Δεύτερη παρατήρηση, ίσως πέρυσι πράγματι δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι έγιναν λιγότερα πράγματα. Ακούστηκαν πολλές κριτικές. Δεν συμφωνώ όμω απόλυτα με τον David Nichols. Δεν συμφωνώ καθόλου με τον David Nichols όταν λέει ότι υπήρξε μια χειροτέρευση. Εμείς είχαμε προσπαθήσει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες που έλεγαν minimum business continuity. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο εκεί όπου δεν έγινε ορατό, σαν τακτική, προσπαθήσαμε να κάνουμε τις απαιτούμενες διορθώσεις. Δεν θέλω εγώ να απολογηθώ ε, για οτιδήποτε άλλον, αλλά παρόλα αυτά δώσαμε κατευθυντήριες γραμμές για όλες τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα τις χρησιμοποιήσουμε και στη Μέση Ανατολή. Υπήρξαν guidebook τα οποία ε, διατυπώθηκαν για τα δικαιώματα των ε, διαφυλετικών προσώπων των ομοφιλοφίλων και των ομοφιλοφίλων σε επίπεδο τοπικών στρατηγικών βέβαια Υπήρξε επίσης μια προσπάθεια την οποία υπενθύμησε ο Νίκολς σχετικά με τον εξορθολογισμό των κατευθυντηρίων γραμμών έτσι ώστε να καταστούν αποτελεσματικότερες και να λειτουργήσουν εκ των κάτω προς τα πάνω. Να ξεκινούν δηλαδή από τοπικές στρατηγικές και δεν τέθηκε θέμα πιλωτικών χωρών. Τώρα υπάρχουν ξεκάθαρες προτάσεις προς τις αντιπροσωπείες στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου χρόνου να αναπτύξουν τοπικές στρατηγικές έτσι ώστε να λειτουργήσουν πιο ελεύθερα οι αντιπροσωπείες αυτές και πιο αποτελεσματικά. Υπήρξε επίσης και το ξεκίνημα της προσπάθειας αναθεώρησης στα ανθρώπινα δικαιώματα, υπήρξε διαβούλευση με εταίρους της κοινωνίας των πολιτών και συζητήσεις με το, Ευρωπαϊκές, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Μπρίζ τον προηγούμενο Απρίλιο στα πλαίσια του ανεπίσημου κοχών. Λοιπόν, τώρα το ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά στον κόσμο, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά υπάρχει μια σχέση ε, ε, αιτία και αιτιατού στη συγκεκριμένη μορφή τη οργάνωση που έχουμε εμεί. Στι επιπτώσει που έχει η οργάνωσή μα και στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου πράγματι γενικά παρατηρεί κανεί ότι τα πράγματα δεν βαίνουν βελτιούμενα. Πώ μπορούμε να οργανωθούμε λοιπόν όπως βλέπετε το οργανόγραμμα είναι μια προσπάθεια της ομάδας Corporate Board της Lady Ashton. Πίσω από όλους αυτούς τους τίτλους αυτό το οποίο είναι σταθερό είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Η πρώτη προσπάθεια δεν είναι μόνο να πληρώσουμε τις θέσεις των λεγόμενων Managing Director. Στα θέματα Global Issues χρησιμοποιεί και τις δύο γλώσσες η, η συγκεκριμένη διευθύντρια η δεύτερη προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε ε, το προσωπικό που έχουμε στη διάθεσή μας, ε, να μην υπάρχουν επικαλύψεις και στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι ώστε να έχουμε το κατελάχιστον θα έλεγα επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού που υπάρχει σήμερα και να τους οργανώσουμε για τη μέγιστη δυνατή, δυνατή αποτελεσματικότητα σε συνεργασία με τον Μπέρτ Τρόιμαν, προς τον οποίο θα μεταφέρω το ιδιαίτερο ε, θετικό μήνυμα το οποίο του απευθύνεται, ο οποίος θα, θα λειτουργήσει σαν, επίσημα σαν πρόεδρος του Κόρουμ στις 25-26 Ιανουαρίου. Βέβαια δεν είμαστε στο ίδιο κτίριο, εγώ θα συνεχίσω ε, να είμαι υπεύθυνη για τις πολυμερείς σχέσεις για ένα χρονικό διάστημα και τα πράγματα γίνονται σε διαφορετικά επίπεδα. Μην θεωρήσετε λοιπόν ότι μέσα σε τρεις εβδομάδες θα υπάρξουν ριζικές αλλαγές. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά τα πράγματα απαιτούν ένα συγκεκριμένο χρονισμό για περαιτέρω συμπληρωματικούς πόρους. Βεβαίως και τους θέλω. Η προτεραιότητά μου δεν είναι να μειώσουμε τα μέσα που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Αν μπορούμε να έχουμε περαιτέρω πόρους, αυτό θα είναι καλό, αλλά δεν θα πρέπει ταυτόχρονα να έχουμε ψευδεστήσεις. Ήταν ήδη πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξουν δύο μονάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεύτερον, αυτό το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη πολιτική σημασία. Αναφερόμαστε ως Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημοκρατίας και ενδώ συνδεόμεθα με το θέμα της εκλογικής παρατήρησης, κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και με τις λεγόμενες πιλωτικές χώρες για τη δημοκρατία και θα συνεχίσω στην αγγλική γλώσσα, λέει η Διευθύντρια. Είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη και εκεί απαιτείται να βελτιωθούν οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας γιατί δεν υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο που ασχολείται με τα θέματα αυτά, στην ουσία δηλαδή μισός υπάλληλος της Επιτροπής και μισός υπάλληλος του Συμβουλίου. Είναι καλό μήνυμα λοιπόν το ότι τέθηκε η λέξη δημοκρατία σε ευρύτερο επίπεδο, σε ευρύτερο τίτλο μάλλον της διεύθυνσης. Τώρα κάποιος ε, που να είναι υπεύθυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Management Board τη υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Φυσικά και αυτό είναι κάτι το χρήσιμο, αλλά δεν ξέρω ποιο θα είναι. Ο Managing Director, αυτό είναι προτεραιότητα της κυρίας Άστον θα έλεγα. θα είναι ένας διπλωμάτης όχι από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, αλλά ένας διπλωμάτης από τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Τέλος, αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία τώρα είναι να διασφαλίσουμε τη διαδραστικότητα στη, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΙΕΣ. Έχουμε αρκετά κείμενα στη διάθεσή μας γύρω από το θέμα αυτό. Πρέπει να διευκρινίσουμε καλύτερα το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της διαχείρισης των οικονομικών ποσών, των ποσών μάλλον που έχει, των πιστώσεων που έχει στη διάθεσή της. Θα υπάρξουν αλλαγές ανάμεσα στην ΤΕΦΚΟ και την ΡΕΛΕΞ, όχι πάρα πολλές αλλαγές, θα πρέπει να συνεργαστούν καλά, τίθενται ορισμένα θέματα για τη συνεργασία και τη συμμετοχή της ΙΕΣ στις οικονομικές δραστηριότητες. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επιληθεί αφού συζητηθεί και ε, ξεπερνά την απλή συνεργασία μας ε, Επιτροπής ΙΕΣ που είναι έτσι και αλλιώς πάρα πολύ καλή. Οι οδηγίες τις οποίες πήραμε το μήνα Οκτώβριο από την Κάθριν Ντέι έλεγαν, ήταν σαφείς, ήταν τόσο σαφείς που δεν ξέρω που τις έχω βάλει. Στην ουσία αυτό το οποίο μας έλεγαν ήταν να συνεχιστούν οι δραστηριότητες ως είχαν, business as usual, και να συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τη Relax όπως το παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι η υπηρεσία αυτή εξωτερικής δράσης δεν είναι μόνο σημαντική σε επίπεδο και πα, αλλά πρέπει να συνεργάζεται στενά με όλους τους συναδέλφους. Φυσικά και εδώ τίθεται θέμα στενής συνεργασία ανάμεσα στις, στα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στις κυριαρχές θέσεις. Και το πολιτικό μήνυμα το οποίο έχει σταλεί στα τέλη Οκτωβρίου είναι διασφάλιση της συνέχειας, συλλογικότητα, ε, συνεκτικότητα στην εξωτερική δράση μας στενότερη συνεργασία προς δύο κατευθύνσεις ανταλλαγή πληροφοριών ίσως και με τον ίδιο τρόπο που γινόταν αυτό ανάμεσα στις διάφορες γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο παρελθόν. Συνεπώς, εσείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ε, παρέχετε τις ε, δικές σας θα έλεγα υπηρεσίες πολλές φορές και με διαιτητικό τρόπο όπως το κάνατε και στο παρελθόν. Είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν συζητάμε τα θέματα των θεωρήσεων ή την μετανάστευση είναι σημαντικό να προσκαλούμε συγκεκριμένα πρόσωπα και να μας προσκαλείτε και εμάς αλλά εσείς θα αποφασίζετε φυσικά ποιοι είναι οι προτιμότεροι για τέτοιου είδους συμμετοχές σε συζητήσεις. Μια τελευταία παρατήρηση αφορά τις αντιπροσωπίες. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το θέμα αυτό. Το θέμα της εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτόπου ε, εξαρτάται κατά πολύ από την αντιπροσωπεία επιτόπου όλα βρίσκονται στα χέρια του, του υπεύθυνου της αντιπροσωπείας, ο οποίος έχει την δυνατότητα να εκπροσωπεί όλες τις αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης σχετικά με την ΚΙΠΑ. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα της εντολής, σε σχέση με την εκπαίδευση των προσώπων αυτών, όπως σας είχε πει η Βαρονιά στις 16 Δεκεμβρίου, έχει δώσει οδηγίες έτσι ώστε όλοι οι νέοι υπεύθυνοι για τις αντιπροσωπείες αυτές να εκπαιδευτούν σωστά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Προσπαθούμε λοιπόν να καθορίσουμε έναν πιο συστηματικό τρόπο εκπαίδευσης. Θα αυξήσουμε φυσικά και την ποσότητα των εκπροσώπων μας στα λεγόμενα σημεία focal points, και έχουμε ήδη σωρεύσει αρκετά καλή εμπειρογνωμοσύνη στο συγκεκριμένο τομέα από συγκεκριμένα κράτη-μέλη για τα λεγόμενα focal points. Οι αριθμοί δεν είναι καθόλου μα καθόλου αρνητικοί. Έχουμε 137 αντιπροσωπείες και έχουμε focal points για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε 120 από αυτές. Και όταν εγώ μιλούσα για 127 μιλούσα για τις επίσημες αντιπροσωπίες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει η κατάσταση είναι αρκετά ικανοποιητική. Αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ένα μια κάποια μορφή δικτύου θα έλεγα Θα πρέπει να καθορίσουμε σωστά το ρόλο τους έτσι ώστε να μην καλύπτονται μόνο από προσωρινούς υπαλλήλου, να μην είναι πάντα κατώτεροι εν πάση περιπτώσει υπάλληλοι ή να έχουν ένα μέντορα στην ιεραρχία προς τα πάνω. Θα πρέπει λοιπόν νομίζω να υπάρξει ένα φόρουμ για όλους αυτούς έτσι ώστε να τους δίνουμε τις σωστές πληροφορίες, να μοιραζόμαστε μαζί τους τις σωστές πληροφορίες και να υπάρχει σωστή ενημέρωση Βέβαια πολλά μένει να γίνουν ακόμα προς την κατεύθυνση αυτή και πράγματι υποφέρουμε αυτή τη στιγμή από έλλειψη πόρων. Φαίνεται ότι έχουν ξεπεραστεί οι δυνατότητές μας και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε παρά να εξετάσουμε. Για την περαιτέρω πρόοδο της παρέμβασής μας, το θέμα της εμπειρογνωμοσύνης και τη συνεργασία όλων των συναδέλφων στα πλαίσια της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης είναι μια πρώτη μάχη που δώσατε και νικήσατε. Η Άστον έχει θέσει τις δικές της προκλήσεις, το λεγόμενο mainstreaming καταρχάς. Θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσουν γεωγραφικά όλες αυτές οι διευθύνσεις και πώς θα υπάρξει επίσης και σωστή ε, πολιτική εκπροσώπωση, γιατί θα πρέπει να υπάρξουν εγγυήσει για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών αυτών. Είπε η Άστον ότι η πολιτική που θα ακολουθήσουμε στον συγκεκριμένο τομέα θέλει να κάνει τη διαφορά. Αυτό συνδέεται για μια ακόμη φορά με την αναθεώρηση. Δεν μπορώ να σας πω πώς θα προχωρήσει η αναθεώρηση. Η τον ενδιαφέρεται περισσότερο με τη δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος, ενός αποτελεσματικού συστήματος και όχι με ένα μικρό ή μεγάλο τελικό κείμενο. Θα απαιτηθεί λοιπόν κάποιος χρόνος, περαιτέρω συζητήσει, συγκεκριμένες αλλαγές βέβαια και σε συνεργασία με την Ίνα και σε συνεργασία με τον Μπέρτο, τον οποίον ενθυμίστε από την Αυστριακή Προεδρία και είναι ένα πρόσωπο ιδιαίτερο σεβαστό στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει επίσης να δούμε και πώς εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εσείς μάλλον, να βοηθήσετε αφού έχουμε εντοπίσει τους συγκεκριμένους τομείς τους οποίους πρέπει να εργαστούμε. Απευθύνω έκκληση όμως για να υπάρξει περαιτέρω χρόνο στη διάθεσή μας. Δεν προσπαθώ να κολυσιεργήσω, αλλά δημιουργούμε νέες δομές. Οι δομές εξαρτώνται από τις νέες πολιτικές πώς θα οργανώσουμε τις πολυμερείς δράσεις μας σε σχέση με τις διμερείς δράσεις, πώς θα οργανώσουμε τις μορφές συντονισμού που είναι ένα θέμα σημαντικό στη διάρθρωση των σχέσεων Επιτροπής και ε, Εξωτερικής Δράσης. Δεν έχουμε ξεκαθαρίσει εντελώς τα πράγματα και πώς οι προτεραιότητες αυτές ε, θα προωθηθούν. Υπάρχουν πολλά θέματα στον τομέα του ανθρωπιστικού δικαίου, σαν παράδειγμα δεν έχουμε κάνει πολλά. Ε, πώς θα συζητήσουμε τα θέματα των διεθνών δικαστηρίων. Προς το παρόν υπάρχει μια διασπορά θα έλεγα των σχέσεών μας με τα δικαστήρια και στο ίδιο το Συμβούλιο. Λοιπόν αυτά με την δική σας βοήθεια, με την εμπειρογνωμοσύνη όλων των συναδέλφων και ελπίζω και με το δικό μου δυναμισμό θα βελτιωθούμε χωρίς αμφιβολία. Α ξέχασα. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι το θέμα αυτό δεν αφορά την πολιτική μας από εδώ και πέρα, αλλά η υπηρεσία αυτή εξωτερικής πολιτικής ελπίζουμε ε, να αποκτήσει μια, ένα νέο εν περιπτώσει όνομα γιατί στα αγγλικά το αρκτικό δεν είναι πολύ κολακευτικό Δεν νομίζω ότι θα είμαστε στο ίδιο κτίριο με αυτούς μέχρι το επόμενο καλοκαίρι τουλάχιστον. Αυτοί που ασχολούνται με την εξωτερική πολιτική θα συνεργαστούν με την κυρία Άστον. Ε, θυμίζω ότι η Άστον είναι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα έχουν αποσπαστεί από τους μηχανισμούς βοήθειας και όλοι αυτοί καλούνται να βοηθήσουν τα θέματα παρατήρησης εκλογών, παρέμβασης πριν από τις κρίσεις, προληπτικές παρεμβάσεις, διορθωτικές παρεμβάσεις κτλ. Και όλα αυτά για μένα και τη διεύθυνσή μου είναι πολύ σημαντικά. Σας ευχαριστούμε για τις ειλικρινείς και ενημερωτικές απαντήσεις σας. Να σας δώσουμε βέβαια κάποιο χρόνο να οργανωθείτε, να εγκατασταθείτε, να οργανώσετε τη συνεργασία με τα άλλα τμήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βέβαια σε αυτό το διάστημα θα είμαστε σε επαφή, θα βλέπουμε πώς προχωρείτε. Τώρα δύο συνάδελφοί μου έχουν ζητήσει τον λόγο, Χάουιτ και Λόχ Μπίλερ. Χάουιτ. Ευχαριστώ. Όπως είπε η κυρία Αρνό, έχουμε κατ' επανάληψη τοποθετηθεί για το θέμα αυτό. Χαίρομαι για την ε, υποστήριξη που έχουμε δώσει στην ε, κυρία Άστον. Χαίρομαι για το διορισμό της κυρίας Αρνό, προσώπου με ιδιαίτερα προσόντα και για το ιδιαίτερο αίσθημα ελευθερίας που διαθέτει. με που λέτε ότι οι τρει εβδομάδε δεν σα φτάνουν για να εκπλώσετε τα καθήκοντά σα, διότι με τα προσόντα που διαθέτετε και τα χαρίσματά σα, είμαι βέβαιο ότι θα ε, επιτύχετε πολλά. Συμφωνώ με τα όσα είπατε για την απαραίτητη εκπαίδευση και αυτά που επικοινωνήσατε είναι σωστά. Εμεί θέλουμε βέβαια σε βάθο εκπαίδευση, είμαι βέβαιο ότι και εσεί το επιθυμείτε, αλλά είναι σωστό και να το πούμε σήμερα. Και το θέμα της στρατηγικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σωστά και αυτά που είπαν προηγουμένως άλλοι παρεμβάντες. Πρέπει να γίνει ορατή και να δημοσιευθεί αυτή η ίσως και να γίνει μια δημοσίευση της στρατηγικής αυτής για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να περιλάβει ίσως και τα συμπεράσματα του ε, Συμβουλίου ε, Υπουργών για τα ε, Υπουργών Εξωτερικών δηλαδή και όλα αυτά να περιληφθούν σε ένα έγγραφο το οποίο θα διανεμηθεί και θα διαβιβαστεί καθώς και με, όπως πρότεινε και ο κύριος Νίκολς. Τώρα, ορισμένα πράγματα με τα οποία δεν συμφωνώ. Κατανοώ ότι για το Συμβούλιο, για το Διοικητικό Συμβούλιο δηλαδή, θα χρειαστείτε κάποιο χρόνο. Αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει μια κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή και η περιγραφή καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα θα πρέπει να τα περιλαμβάνει τα πράγματα αυτά και να διαθέτει βέβαια νομική παιδεία ο αρμόδιος αυτός αξιωματούχος. Πρέπει να συνεχίσουν να πιέζουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Σε ό,τι αφορά τα σημεία εστιασμού, είναι ένα θέμα το οποίο τέθηκε στη συζήτηση. Ο προγραμματισμός του EHDR έχει γίνει και στο παρελθόν πάλι από πρόσωπα με νομική παιδεία. Ο κίνδυνος που υπάρχει είναι ότι αν το διευρύνουμε ίσως να υπάρξει κάποια αποδυνάμωση των ικανοτήτων των αρμοδίων αξιωματούχων. Ίσως δεν έχω λύση να σας προτείνω τώρα, αλλά πρέπει να είναι ένα θέμα το οποίο ψάσουμε. Για το θέμα των αριθμών που σωστά έθεσε ο κύριος Νίκολς. Για το θέμα των αριθμών. Είναι βέβαια δύσκολο και είναι και είμαστε και σε περίοδο οικονομικής στενότητας. Αλλά δεν είναι θέμα στο οποίο επίπεδο θα κινηθούμε. Θέμα απόδοσης περισσότερο. Όπως είπαν όλοι, υπήρξε επιδίνωση το προηγούμενο χρόνο. Δεν γνωρίζω αυτό είναι σωστό ή όχι. Αλλά δεν θα, υπάρξει, δεν θα πρέπει να υπάρχει επιδίνωση σε σχέση με το παρελθόν να φροντίσουμε να υπάρχουν οι απαραίτητες δυνατότητες. Γνωρίζουμε ότι η Προεδρία έχει φέρει τις ικανότητες αυτές και στις Βρυξέλλες και στην Γενέβη, τους πόρους αυτούς. Τις ίδιες ικανότητες θα πρέπει να διατηρήσουμε λοιπόν και για το μέλλον. Αυτό μας ζητούν και οι ε, μη κρατικέ οργανώσεις και αυτό το μέτρο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την διαρκή έδρα του co Home τώρα θα είμαι λίγο ριζοσπαστικότερος. Είναι σωστό να υπάρχουν ανώτεροι οξωματούχοι από τις πρωτεύουσε για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και να υπάρχει συνεργασία μαζί τους και είναι καλύτερο αυτό παρά να υπάρχει μια μόνιμη έδρα στις Βρυξέλλες όπου τότε οι αξιωματούχοι που θα βρίσκονται μονίμως εδώ θα έχουν λιγότερη επιρροή στις πρωτεύουσε. προσωπικά προτιμώ μια μόνιμη έδρα του Κόχομ στις ε, Βρυξέλλες. Αλλά ε, βλέπω αυτή την δυσκολία. Ε, εν τέλει, για το θέμα αυτό του mainstreaming, να γίνει συζήτηση με τους συναδέλφους μας της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων. Η κυρία Αρνό έχει δίκιο που τα λέει αυτά δεν μπορεί να γίνει mainstreaming χωρίς την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη. Θα πρέπει να εκπαιδευτούν ορισμένοι της EAS για τις βασικές αυτές αρχές. Χρειαζόμαστε ανθρώπους όπως η κυρία Αρνό που να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις, να σχολιάζουν τα έγγραφα, να διαβιβάζουν πληροφορίες. Και αυτό πρέπει να το προωθήσουμε και να γίνει μια συζήτηση μεταξύ κοινοβουλίων και άλλων ε, αρμόδιων θεσμικών οργάνων. Η μέθοδος εργασίας θα πρέπει να είναι η ίδια όπως με θέματα εμπορίου και ανάπτυξης. Θα πρέπει να βελτιωθούν και οι προσδοκίες του Κοινοβουλίου. Εάν θέλουμε δηλαδή η EEAS, η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων, να αρθεί στο ύψο των προσδοκιών μας, θα πρέπει τα αρθρόπαιτα δικαιώματα να παίξουν σημαντικότερο ρόλο σε όλες τις πολιτικές και τι εμπορικέ πολιτικέ. Και αυτό που πρέπει να απασχολήσει το Κοινοβούλιο είναι κατά πόσον και με ποιου μηχανισμούς. Συγχαίρω και πάλι για τον διορισμό της την κυρία Αρνό και ευχαριστώ και τους άλλους παρεμβάντες για τις ε, παρεμβάσεις τους. Ευχαριστώ για τις ε, παρατηρήσεις σας, αγαπητέ Ρίτσαρντ. Η κυρία Λόχ Μπίλερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα γερμανικά, που είναι και η μητρική μου γλώσσα. Ο Ρίτσαρντ Χάουιτ είπε πολλά για λεπτομέρειε. Εγώ θα έρθω σε ορισμένα συγκεκριμένα μόνο θέματα. Απευθυνόμενη πρώτα σε εσά, κυρία Αρνό, σα εκφράζω τα συγχαρητήριά μου για τον διορισμό σα και εμεί οι πράσινοι σας ακούσαμε στην εσωτερική μας ακρόαση και σας βρήκαμε και γνώστρια του θέματος και δυναμική. Θυμούμε τώρα τη συζήτηση που κάναμε στην Ολομέλεια του Στρασβούργου με την Λέβη Άστον, όπου ένα θεμελιώδες θέμα της συζητήσεως αυτής ήταν το mainstreaming και βεβαίως το υποστηρίζουμε. Όμως από μόνο του, εάν μείνει μόνο το αυτό το mainstreaming θα αποτελέσει οπισθοδρόμηση δεν έχουμε ακόμα την βεβαιότητα ότι θα υπάρξει διεύθυνση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα για το τρίτο θέμα που περιλαμβάνεται στο ψήφισμά μας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι θέλουμε δηλαδή υψηλού επίπεδου προσωπικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδική εισηγήτρια, ειδικό εισηγητή ή εκπρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι μια αξίωση που έχει ε, υποβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που έχει υποστηριχθεί και ιδίω από τη δική μα πολιτική ομάδα. Είναι θέμα βεβαίω ικανότητα σε όλα τα επίπεδα. Την τελευταία φορά στην Νομική Επιτροπή ρώτησα τον εκπρόσωπο της Βελγικής Προεδρίας ποια είναι τα κυρίαρχα θέματα της Ουγγρικής Προεδρίας και μου απάντησε ότι δεν χρειάζεται να ρωτάτε τι θα γίνει, θα τα κάνει αυτά στο μέλλον η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. βρισκόμαστε τώρα σε μεταβατική περίοδο. Υπάρχει ωστόσο πρόβλημα ικανότητα με την έννοια της capacity δηλαδή. Και η εκπροσώπηση η εκπροσώπηση το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίδραση για το θέμα της θυνησίας από την κυρία Άστον είναι άξιο επικρίσεων ο θέμα τώρα των αντιπροσωπιών, μιλήσατε πριν, ε, μιλώντας για focal points για τους ε, υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, είπατε ότι ορισμένε ε, αντιπροσωπίες είναι πάρα πολύ περιορισμένες, πολύ μικρές. Όμως υπάρχουν 120 αντιπροσωπίες που έχουν τέτοιες αρμοδιότητες μέσα στα πλαίσια της Ένωσης και μέσα σε, στην Ένωση αλλά και μέσα σε πολυμερή όργανα. Δεν μιλώ εδώ για τις πολύ μικρές εκπροσωπήσεις. Ένα μεγάλο μέρος των αντιπροσωπιών αυτών έχουν focal point που μπορεί να εργαστεί 100% για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και εκδημοκρατισμού. Καμιά φορά οι αξιωματούχοι αυτοί είναι πολύ junior, δεν είναι δηλαδή ε, σε αρκετά υψηλέ θέσεις. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν έχουν, ε, δεν έχουν επαρκή προσόντα. Αλλά ε, βρίσκονται, είναι χαμηλόβαθμοι δηλαδή στις πρεσβείες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Οι προσδοκίες τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων έχουν αυξηθεί και πιέζει μεν ο χρόνος αλλά όταν ρωτούμε μας απαντούν διαρκώς ότι όλα αυτά βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο, στο στάδιο των, ε, ε, της επεξεργασίας. Αυτά δεν έχουν καλά προς τα έξω. Βεβαίω και πρέπει να καταπολεμήσουμε τα διπλά μέτρα και σταθμά, αλλά να το κάνουμε αυτό και μέσα στο ίδιο το κοινοβούλιο. Διότι έχουμε την κατάσταση όπου επικρίνουμε σε ψηφίσματά μας και τα περνάμε εύκολα τα ψηφίσματα αυτά ως επίγοντα κλπ. Για ορισμένες χώρες, αλλού όμως για άλλες χώρες όχι. Αυτά δεν μπορούμε να τα φορτώνουμε λοιπόν όλα στις πλάτες της υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Μάλιστα, λέει κυρία Χάουταλα. Να εξετάσουμε όλοι λοιπόν πώς ε, μπορούμε να είμαστε κάπως συνεκτικότεροι στο πώς χειριζόμαστε τα θέματα των διαφόρων χωρών. Δεν βλέπω να ζητούν άλλοι το λόγο, επομένω ήρθε η ώρα ο Ντέιβ Νίκολ να απαντήσει. Ε, η κυρία Αρνό. Κοιτάξτε, έχουμε άλλα δύο θέματα σήμερα στη διάταξη. Ντέιβ, όμω έχει πρώτο το λόγο. Πάρα πολύ σύντομα θα σα τα πω για να επανέλθω ει κάποια από τα σημεία τα οποία ανέφεραν και όσον αναφορά τα προβλήματα του 2010. Δεν θέλω να το παρακάνουμε. Απλώς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναγίνουν αυτά όσο προχωρούμε με τη νέα διάρθρωση. Δυστυχώ τα πράγματα είχαν εξαιρετικό χαρακτήρα. Πέρσι δεν ήταν συνείδηση πρώτων πραγμάτων και άρα θα κάτσουμε να δούμε τι συμπεράσματα ελήφθησαν, τι ελέγχθη όσον αφορά τι ατομικέ επισκέψει σε κάποιε χώρε και να διαπιστώσουμε τι θα έπρεπε να περιμένουμε να γίνει και που δεν θα γίνουν. Επίσης να βρω κάποιες ε, δηλώσεις γιατί η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν η γλώσσα του δικαίου τροπίνου δικαιωμάτων, ήταν περισσότερο γλώσσα της γεωπολιτικής, της γεωστρατηγικής και των αντιστοίχων διεθνών σχέσεων, το οποίο πάνε να πει ότι αυτοί που είχαν την εμπειρογνωμοσύνη για δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διεθνέ δίκαιο κλπ. δεν ενεπλάγησαν ή δεν ήρθε υπόψη γνώμη του και. Έρχομαι σε κάτι άλλο για την Τινησία. Δυστυχώ είναι μία από τι πολλέ περιπτώσει κατά τι οποίε δεν είναι απλά θέμα δυνατοτήτων η έλλειψη αυτών που οδηγούν εις αδράνεια είναι περίπτωση απουσίας πολιτικής βούληση. που δεν μπόρεσε ε, ε, κάτι το οποίο πρέσβευε κάποιος να το προωθήσει. Γιατί δεν θέλουμε τα κρατη Τώρα έχει η θέση μας αποδυναμωθεί. Θα μπορέσει τώρα η υπηρεσία εξωτερικής δράσης να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει τώρα. Όσον αφορά την Κόχομ στις Βρυξέλλες, Εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν γραφεία στις πρωτεύουσε. Θα συνεχίσουν να έρχονται οι εμπειρογνώμονες οι ειδικοί από εκεί εδώ. Και εδώ η υπηρεσία θα προσθεθεί στο οργανόγραμμα. Και θα πρέπει αυτής εξ αρχής να ξεκαθαρίσουμε τι εντολή θα έχει η υπηρεσία των Βρυξελών σε σχέση με τις κατατόπους τι ύλη θα πρέπει να και λοιπά Να παρακολουθεί όλη την εξωτερική πολιτική, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Κάποιοι από τους ειδικού ε, αφού είναι στους ε, πρωτεύουσες να το παρακολουθούν. Όλα αυτά οι συνάδελφοι ας πούμε που δουλεύουν ας πούμε για το Μαγκρέβ μπορούν να ξέρουν τι λέει η Ευρώπη για το Μαγκρέβ δηλαδή για την προσωπίες. Όντως θέλουν περισσότερους πόρους. Και γι' αυτό και έχουμε υποβάθμιση της δουλειάς τα τελευταία χρόνια. Και οδηγηθήκαμε σε σύγχυση. Και στο παρελθόν είχαμε πρεσβείες που είχαν θετική στάση και τώρα μου τους απευθυνθεί κάποιος εκεί, τον στέλνουν στην προσωπία της Ένωσης. Να ξεκαθαριστεί στα κράτη-μέλη όμως ποια είναι η ευθύνη τους. Γιατί οι προσωπίες επλήγησαν και θα συνεχίσουν να πλήσονται από το ότι τώρα υπάρχουν λιγότεροι πόροι. Ε, να βρεθούν πιο δημιουργικοί τρόποι, ούτως ώστε να βοηθήσουν κάποιοι ειδικοί, πρεσβείες. Χρειάζεται περισσότερη ευελιξία. Και έτσι να μπορούν τα κρατημέλη, εκεί που υπάρχουν κάποιοι που ξέρουν επιτόπου να βοηθούν. Αυτά. Thank you very much, Dave. Uh, now... Dave, σε ευχαριστούμε. Βερονίκ, μήπως θέλεις να μας πεις και εσύ κάτι. Βερονίκ. Έχει δίκιο ο κύριος Νίκολς εκεί που λέει για το ότι υπήρχε άλλη γλώσσα. Δεν υπήρχε τέτοιο είδους timing, χρονισμός που μας οδηγεί να τα χαρακτηρίσουμε αυτά παιδικές ασθένειες υπηρεσίες. Αυτά τα, τα ψηφίσματα όλα που βγήκαν ε, συναντήσεις με Ιράν, με Καναδά, με Βόρεια, Κορέα. Ναι, ναι, καλά δεν όλα, αλλά συμφωνώ ότι είχαμε κάποια θέματάκια εκεί. Όχι για την Τινησία δεν με μεγάλη μου χαρά διαπίστωσα ότι ήταν πάρα πολύ αποφασιστικός ο εκπρόσωπος σήμερα το πρωί, εκπρόσωπος της Άστον Και εμεί προσχωρούμε στην με ανθρωπινά και δημοκρατία βλέπουμε ότι είναι σαφή η σχέση μεταξύ ανθρωπινών δικαιωμάτων και του πώ εξελίσσεται η κατάσταση. Γιατί χρειάζεται αναβάθμιση των διμερών σχέσεων. Οπότε δεν ξέρω για τους άλλους, αλλά σήμερα το πρωί ο εκπρόσωπος της Άστον τα είπε έξω τα δόντια για τις υπηρεσίες, για την κοχόμ, για την υποβάθμιση των προσωπιών, τα άκουσα και το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσουν να κρατημένα να θεωρούν ότι είναι συνυπεύθυνα, δεν θέλουμε άπαξ. Και την προσωπία θεωρεί ότι έχει λόγο στην συντονισμό να κατεβάζει τον πύχη όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με το παρελθόν. Γιατί παλιότερα οι την ήταν η φωνή της Ένωσης. Και αυτό που είπε ο Ντέβιντ, ότι σε κάποιες περιπτώσεις ε, πήγαινε, στενόταν κάποιος από τον Άννα στον Καϊάφα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ καλή η εμπειρία, η γνώση που υπάρχει στις, στις Είναι κρίμα να πάει. Να χαθεί. Ροή τη πληροφοριών. Δεν θέλουμε τα κράτη-μέλη να θεωρήσουν ότι πια ξέφυγε από τα χέρια του η υπόθεση. Φυσικά και είναι δική του υπόθεση. Λόγω των κρατομελών έχουμε εξωτερική πολιτική, έχουμε θεωρήσει διαβατηρίων, όλα αυτά που έχουμε. Χάρη σε αυτά, τα κρατη μπορούμε να έχουμε την υπηρεσία και το διπλωματικό σώμα. Δεν θα τα καταφέραμε χωρίς τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται πάντως και από τις δύο πλευρές καλή διάθεση. Ε, αυτό που είπα τώρα για την προσωπικότητα. Πέρσι το είχε πει η κυρία Στον, ότι είχαμε κάπως πλεόνασμα. Να δούμε πώς θα δημορφωθεί η κατάσταση και να καταλήξουμε κάπου μέχρι 3 Φεβρουαρίου, γιατί ακριβώς θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την εντολή που θα διέπει τους ειδικού εκπροσώπους της Ένωσης που τον οποίο εντολή εκπνέει. Πάντως θεωρώ ότι δεν πάμε προς τα εκεί. Μάλλον πάμε προς το να έχουμε μια ολόκληρη ιεραρχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα προς το παρόν ο Πιέρ είναι ο αρμόδιος δεν ξέρω θα κάνει στο μέλλον Αυτά σε υψηλό επίπεδο. Αυτά, αυτά ήθελα να σας πω. Και βεβαίω ευχαρίστω να συνεχίσω να σας ενημερώνω, να ακούω τις ιδέες σας, γιατί η επιτυχία είναι στόχος και ημών και ημών. Εμείς ευχαριστούμε λέει πρόεδρος και ευχαριστούμε και εσένα και τον πρόεδρο θα συνεχιστεί η συζήτηση. Και τώρα. Και τώρα έχουμε τον πρόεδρο της Υποπιτροπής μας, ο οποίος θα πάρει την σκητάλη, γιατί ξέρετε, Έχω jet lag ήταν το ταξίδι που μου έχει τσακίσει από τη Μαλαισία. Θα πρέπει να κάνω μια βολτίτσα, αλλά δεν θα την κοπανίσω. Για λίγο θα προεδρεύσει ο Άντρε. Άντρε, έχεις το λόγο. Πρόεδρε, Σας εύχομαι να ξεκουραστείτε. Περνάμε στο 6 τώρα, τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Εξωτερικών Συνόρων Frontex. Έχουν υπάρξει ορισμένες τροπολογίες οι οποίες έχουν ήδη κατατεθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά αυτή την έκθεση, έχουμε τις ημερομηνίε 25 και 26 Ιανουαρίου. Και, και η Άφετ, αλλά και η Ντρουά, θα πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας για το θέμα. Πρώτα πρώτα όμως να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή κύριο Λόχμπιλερο γιατί ήταν ε, ο συντάκτης έκθεσης, ε, της εκθέσεως η οποία προσέστηκε πρώτη φορά στις 14 Δεκάτου στην Επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, είχε γίνει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, παρουσία μη κυβερνικών οργανισμών, διαφόρων φορέων, παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης ε, έχουμε νέα τροπολογίες οι οποίες έχουν υποβληθεί, συμβιβαστικές τροπολογίες. Εκτός από τις ε, αρχικά υποβληθήσεις, 44 από διαφόρους συναδέλφους ευρωβουλευτές. Και λόγω της εξαιρετικής συνεργασίας καταφέραμε να καλύψουμε όλες τις ε, προσδοκίες σας. Ότι, ζητήσατε δηλαδή στις τροπολογίες. Οι, οι σκιώδες ηγητές προέρχονται από όλες τις ε, πολιτικές ομάδες Όλε, όλες τις πολιτικές ομάδες και φαντάζομαι θέλουν το λόγο. Κυρία Λόχμπιλερ. Κυρία, κυρία Λόχμπιλερ, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντα την νομική υπηρεσία και ε, το Κοινοβούλιο που μας βοήθησαν με αυτήν την ε, έκθεση. Ήταν πολύτιμη η βοήθειά τους. Να μην τώρα αναλύσω μία-μία τροπολογία, αλλά ο σκοπός της η υπηρεσίε μα είναι η Frontex να λαμβάνει περισσότερη υπόψη τα ανθρωπινά δικαιώματα, να τα σέβεται για τι σχετικέ αρχέ του δικαίου των ανθρωπινών δικαιωμάτων και ότι έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε τη δουλειά τη Frontex να γίνει πιο αποτελεσματική. Να μπορούμε να έχουμε ψηλότερα τον πύχη για τα ανθρωπινά δικαιώματα από ότι προηγουμένω. Επομένω έχουμε μία αξιολόγηση αμερόληπτη ανεξάρτητη και περισσότερη διαφάνεια από τη Frontex όσον αφορά τις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προφορικά για να υπάρχει τακτική ενημέρωση και γι' αυτό σας λέω θέλουμε να υπάρχει ακριβής διατύπωση στην έκθεση για το πώς θα τηρούνται τα προβλήματα από το διεθνές δίκαιο, από το δίκαιο δικαιωμάτων, να μην είναι γενικόλογες οι διατάξεις. Να ενθαρρυνθεί η Frontex να χρησιμοποιήσει εμπειρία, γνώση των διεθνών φορέων όπως της Πατσαρμοστίας, όπως ε, της Επιτροπής των Δικαιωμάτων και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει σχετική κατάρτιση που δεν έχει γίνει πριν, κατάρτιση για ανθρώπινα δικαιώματα και για να δούμε την... το περιεχόμενο τώρα. Πρόκειται για την δεύτερη φορά που τα συζητάμε αυτά στην Επιτροπή μας. Ξέρετε, την τελευταία εβδομάδα πριν το Στρασβούργο είχαμε μια σειρά διμερών συναντήσεων με τους σχεδόν και με άλλα μέλη του Κοινοβουλίου. Και μέχρι σήμερα το πρωί εγώ επρέσβευα το ότι μπορούμε να βρούμε συμβασμό. Αλλά τώρα την ώρα της συνεδρίασης θεωρώ ότι η η συμβαστική 7 δεν μπορεί να παραμείνει. Γιατί τελικά υπήρξε απόκληση από των απόψεων αυτών που στην αρχή συνεφώνησαν επίσης όσον αφορά τις αρχικές μου. Ο κ. Κομοτσάκος της Λίμπε που είναι ο σκιώδη ηγητής του ΕΛΚ και εκείνος είπε ότι αμφισβητεί κάποιες από τις προτάσεις μου. Ίσως σε κάποια σημεία μπορέσουμε να τα βρούμε, άλλωστε πρόκειται για μεγάλο κατάλογο θεμάτων, αλλά για όλα θα δυσκολευτούμε. Καλά, ίσως θα πρέπει να μας πείτε και, εσείς, ο ίδιος τη γνώμη Έχουμε όλες αυτές τις συμβαστικές, είπαμε, οι οποίες ελπίζω ότι θα ισχύσουν και έχουμε και δύο προφορικές. Ζήτησα από τους συναδέλφους να μου πούνε αν δέχονται το συμβασμό. Να μου πούνε. Δύο γενικές παρατηρήσεις τώρα. Τροπολογίες που αφορούν τον εισηγητή του ΕΛΚ, τον κύριο Κουμουτσέκο. Ε, πρόκειτο όχι για θέματα στενά ειδωμένα των δικαιωμάτων. Πολλές αυτές τις τροπολογίες σχετίζονται με, για τη σχέση μεταξύ Frontex και εθνικών κυβερνήσεων. Όμως δεν έχουμε εδώ άλλες ε, επιτροπές, οπότε του είπα ότι καταρχήν εντάξει θα συμπεριλάβω τα όσα πρότεινε ή στο σχέδιο κειμένου μου και ε, θα τα συζητήσουμε ελπίζω ξανά εδώ και να δούμε τι γίνεται με κατροπολογίες που νομίζω ότι ε, τελικά δεν έχει κανείς ένσταση, τα είπαμε το Δεκέμβριο, όμως σε όλο αυτό το έγγραφο δεν σημαίνει πουθενά η έκφραση παράνομος. Λέμε παράτυπος ή αντικανονικός. Και τα είπαμε και στη Βαρσοβία. Αυτό. Το αντικανονικός είναι πιο δοκιμός όρος. Το είπε και ο επικεφαλής της ε, της Frontex. Η ήδη, αυτό επομένως μπήκε στο κείμενο, θεωρώντας ότι θα περάσει αυτή η διόρθωση εις όλο το κείμενο. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά από τα όσα μεταφράστηκαν. Θα τα ψηφίσουμε όλα αυτά στην ΑΦΕΤ την Πέμπτη. Σας ευχαριστώ. Ήθελα να σε ρωτήσω αν κάποιος επιθυμεί να λάβει το λόγο για τις προτάσεις αυτές. Ξεκινώντας αμέσως την κυρία Λόχμπιλε για την ε, συνεργασία που πράγματι είχαμε, αναλυτική συνεργασία για μια σειρά σημείων ε, του κειμένου που συζητάμε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι το κείμενο για την ε, τροποποίηση του κανονισμού της Frontex είναι ένα σημαντικό κείμενο. Και από νομοθετικής και από πολιτικής πλευράς. Όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση, ο βασικός σκοπός είναι να συνθέσουμε δύο πράγματα. Αποσκοπούμε στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και της αποτελεσματικότητας της Frontex, διασφαλίζοντας και προάγοντας ταυτόχρονα τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η οθέτηση λοιπόν ενός τόσο σοβαρού κειμένου θα έχει άμεσες και χειροπιαστές συνέπειες και αντίκτυπο στην κοινή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αλλά και σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες μας το πολύπλοκο και δύσκολο πρόβλημα της αυξημένης παράνομης ή παράτυπης μετανάστευσης προς την Ευρώπη. Νομίζω και εδώ θα ήθελα να, το, να αναφερθώ σε αυτό πολύ σύντομα. Νομίζω ότι είναι περιττό να κάνω αναφορά στην κυριολεκτικά ζωτική σημασία που έχει η αποτελεσματικότητα της Frontex για μια χώρα εταίρο που είναι πραγματικά στο σύνορο της Ευρώπης και αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα στην αντιμετώπιση ενός μεγάλου κύματος παράνομης, παράτυπης ή λαθρέας μετανάστευσης. Το γεγονός ότι είμαι Έλληνας, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί να με κάνει παρά να έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στην αποτελεσματικότητα της Frontex αλλά και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 90% το 90% επαναλαμβάνω των λαθρέων μεταναστών ή των παρανόμων μεταναστών ή των παρατύπων μεταναστών αυτό είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε και να το βρούμε που έρχονται σε ευρωπαϊκό έδαφος το πρώτος, ο πρώτος σταθμός τους είναι η χώρα μου. Επομένως όσο και αν ήθελα δεν μπορούσα παρά να είχα στις προτάσεις και τις τροπολογίες μου υπόψη μου και αυτά τα σκληρά δεδομένα, αυτή, τα δεδομένα αυτής της σκληρής πραγματικότητας. Επομένως, αυτή είναι η λογική και αυτός είναι ο επιδιωκόμενος στόχος των τροπολογιών που υπέβαλα ως σκιώδης εισηγητής για το ΕΛΚ. Δεν κάνω καμία έκπτωση στην ανάγκη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά δεν μπορώ να κάνω και καμία έκπτωση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης Frontex όσον αφορά τις τροπολογίες και τις προτάσεις της εισηγήτριας της κυρίας ε, Λόγμπιλε. Αφού την ξαναευχαριστήσω για τη συνεργασία και το πνεύμα κατανόησης, θέλω να πω ότι έκρινα με ανοιχτό πνεύμα αυτές τις προτάσεις, με πολύ καλή διάθεση και σεβόμενος τις ευαισθησίες που άλλωστε είναι και δικές μου, καθώς και τη σημασία την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπου διαφωνώ, με όποιες προτάσεις της κυρία Λόγμπιλε διαφωνώ, το κάνω μόνο όταν είμαι απολύτως πεπισμένος ότι τυχόν η υιοθέτησή τους θα επιβαρύνει υπερβολικά το μηχανισμό της Frontex με αρνητικές συνέπειες στην επιχειρησιακή της ετοιμότητα χωρίς ταυτόχρονα να επιτυχάνεται μια πραγματικά κρίσιμη προστιθέμενη αξία στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με τα όσα ήδη, προ όσα ήδη προβλέπονται στο κείμενο της Επιτροπής. Μόνο τότε διατυπώνω διαφωνίες αλλά και πάλι το πεδίο συνεργασίας, έστω και αν είναι πολύ κοντά η ψηφοφορία στην ΑΦΕΤ, είναι την επόμενη Πέμπτη, <clears throat> και μέσα σε αυτό το πνεύμα είμαι και πάλι διατεθειμένος να αναζητήσουμε ε, σημεία και κοινού τόπου. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις συγητές καθώς και τους συναδέλφους, μέλη της Επιτροπής για την πολύ καλή δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιθυμεί κανείς άλλος συνάδελφος να λάβει τον λόγο για τα θέματα, για, τα, τις τροπολογίες ή προφορικές τροπολογίες. Κανείς. Α, η κυρία, η κυρία, η Λοχπίλερ. Αν δεν ακούσω από τους κοιόδης συγητές, είτε τους σοσιαλιστές, είτε τους φιλελευθέρους είτε την ΓΚΟΕ θα είναι δύσκολο να κάνω μια σύνοψη διότι τώρα με το feedback το έλαβα μόνο σήμερα βέβαια δεν μπορώ να μιλήσω να πω ποια είναι η θέση των υπολείπων ελπίζω λοιπόν αύριο ή μεθαύριο να έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα δηλαδή πόσο μπορούμε να υποστηρίξουμε τις διάφορες συμβιβαστικές τροπολογίες. Εν τέλει θα ήθελα να πω ότι η πρόθεσή μου βέβαια δεν είναι να βάλω κολλήματα στο έργο της Frontex, αλλά θα εξετάσω όλες τις συμβαστικές τροπολογίες που πηγαίνουν και προς το άλλο άκρο. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό. Να έχουμε δηλαδή εν τέλει ένα έγγραφο το οποίο να λέει ωραία λόγια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς όμως πραγματική πυγμή σε ό,τι αφορά την, την αξιολόγηση, την ε, εξέταση των όσων πράττει η Frontex τότε στην περίπτωση που φτάσουμε σε κάτι τέτοιο θα αποσύρω την υπογραφή μου αλλά ελπίζω δεν θα φτάσουμε σε κάτι τέτοιο Σας ευχαριστώ πολύ ε, κυρία μου ελπίζω ότι θα βρεθεί ε, μια ε, ικανοποιητική λύση ικανοποιητική λύση και <clears throat> είμαι πεπισμένος ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε σε αποφάσεις όπως η απόσυρση της υπογραφής από ένα κείμενο. Είμαι βέβαιος ότι η ικανότητα της κυρία Λογμπίλε θα μας οδηγήσει σε ένα κείμενο συμφωνημένο. Ε, θα ήθελα μόνο να πω, ε, κύριε Πρόεδρε, ότι επιμένω ότι οι όποιες ανησυχίες ή όποιες αντιρρήσεις διατύπωσα αφορούν πραγματικά περιορισμένο αριθμό των προτάσεων και των ε, εισηγήσεων της κυρίας Λοχμπίλε και σας είπα με ποιο, με ποιο λόγο. Από εκεί και πέρα, ε, εμείς σήμερα και αντιλαμβάνομαι ότι ίσως είμαστε οι μόνοι που έχουμε ενημερώσει την κυρία Γλωγομπίλε αναλυτικά για τις θέσεις μας σημείο προς σημείο. Πάνω σε αυτό βεβαίως θα περιμένουμε, αντιλαμβάνομαι την υποχρέωσή της ε, και το λογικό του αιτήματο να περιμένει και αντιδράσει από τι άλλε πολιτικέ ομάδε. Πάντω, εμεί είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και να αναζητήσουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι μετά την δήλωση αυτή η κυρία Λοχμπίλερ θα μπορέσει να αναζητήσει λύσεις σε συνεργασία μαζί σας. Ο κ. Χάουιτ. να ζητήσω συγγνώμη από την κυρία Λόχπιλερ. Θα έρθει σε επαφή με το σκιώδη εισηγητή τις επόμενες μέρες. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, εν πάση περιπτώσει. Σας ευχαριστώ, λέει πάλι ο Νομίζω ότι εδώ μπορεί να λήξει η συζήτηση του υπαριθμών 6. Υπάρχει ακόμη ένα θέμα. Ε, μας μένουν όμως ε, το πολύ 15 λεπτά έχουμε το υπαριθμό 7 έκθεση δηλαδή απολογισμός απολογισμός μάλλον από πλευρά των βουλευτών που συμμετέσχουν στην αντιπροσωπεία της ΑΦΕΤ στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Μια δεκαμελής αντιπροσωπεία η οποία μετέβη εκεί στην οποία συμμετέσχε και η κυρία Λόχ Μπίλερ, η στον Παρόδο, διεξήχθησαν πολλές συναντήσεις στα πλαίσια της μεταβάσεως της αντιπροσωπείας. Εκεί κυρίως συζητήθηκαν θέματα απτόμενα της Αφρικής, των εξελίξεων στην Αφρική, Νότιο Σουδάν. Νομίζω το θέμα του Σουδάν ήταν και το πιο σημαντικό αντικείμενο των συζητήσεων. Αναμένουμε τώρα τα αποτελέσματα του δημοσιοφίσματος του Σουδάν. Η κυρία Λίνε Άντβιτσον του είπα του εκπροσώπου ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι παρούσα εδώ και θα την παρακαλέσω εάν επιθυμεί να ε, κάνει κάποιο σχολιασμό της, της αποστολής αυτής. Έχω βέβαια και τον κύριο Λάιχτφριντ που συμμετείχε στην αντιπροσωπεία και ίσως θα έπρεπε αυτός πρώτος να λάβει το λόγο. στα Είναι κρίμα που έχω μόνο 10 λεπτά γιατί είχα ε, προετοιμαστεί να μιλήσω τουλάχιστον μισή ώρα. Ξεκινώντας, να πω ότι η αντιπροσωπεία παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ήταν σωστά προετοιμασμένη, είχαμε συναντήσεις υψηλού επίπεδου, και από ό,τι φαίνεται οι αλλαγές που προκλήθηκαν από τη συνθήκη της Λισαβόνας μας επηρέασαν στις αντιπροσωπείες μας γιατί έχουμε την δυνατότητα τώρα να συναντώμεθα με ε, ομιλητές υψηλού επίπεδου, συνομιλητές υψηλού επίπεδου. Όπως είπατε και εσείς ε, κύριε Πρόεδρε για την περίπτωση του Σουδάν, αυτό ήταν ένα από τα θέματα τα οποία είχαμε την δυνατότητα ανάμεσα σε άλλα να συζητήσουμε. Όλοι οι εταίροι τους οποίους είχαμε τη δυνατότητα να δούμε είχαν αγωνία για το πώς θα πάει το δημοψήφισμα, για το εάν είναι δυνατό να προετοιμάσει κανείς ένα τέτοιο δημοψήφισμα σε μικρό χρόνο, μια μεγάλη προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών και όλων των υπολείπων εμπλεκομένων και από ό,τι φαίνεται το δημοψήφισμα αυτό πήγε σχετικά καλά, τυπικά τουλάχιστον, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον από τις ανακοινώσεις των τύπων. Το θέμα γενικότερα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χρηματοδότησης. Η οικονομική κρίση φαίνεται παρεμποδίζει τα Ηνωμένα Έθνη να έχει αρκετά χρήματα στη διάθεση του για παρεμβάσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεωρούν ότι τα κράτη-μέλη έχουν λιγότερα χρήματα για τις οργανώσεις όπου η συμμετοχή, η συνδρομή, αν θέλετε, δεν είναι υποχρεωτική. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έχει ε, κάποια προβλήματα στην οργάνωση των υπηρεσιών της ανάμεσα στη Γενέβη και, τα, και τη Νέα Υόρκη και ίσως πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη κατανομή θα έλεγα αρμοδιοτήτων και ε, γενικά ύλης ε, προς εξέταση ανάμεσα στις δύο πόλεις. Ε, μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσης παρέμβαση ήταν ο τρόπος αντιμετώπισης της κατάστασης που υπάρχει σε ορισμένα κράτη-μέλη, τα οποία συμμετέχουν στις εργασίες του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο δεν είναι βέβαια και πάρα πολύ θυμισμένο για ένα τέτοιο σύστημα λειτουργίας έχει νόημα δηλαδή να συμμετέχει κανείς εκεί στο Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για να βοηθήσει ή μήπως είναι προτιμότερο να προσπαθήσει να συνδράμει εκτός. Ένα άλλο, θέμα, ένα άλλο θέμα μάλλον εκτός ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ότι η Ένωση μετά τη Λισαβόνα προσπαθεί στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών να λειτουργήσει με πιο ε, θα έλεγα καθοριστικό τρόπο. και τίθεται το θέμα ποιος εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ποιο επίπεδο και περιέργως όλες αυτές οι χώρες ε, οι οποίες είχαν ψηφίσει πριν μερικές εβδομάδες πριν πάμε εκεί, όλες οι χώρες οι οποίες ε, αντιμετωπίζονται καλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα σε θέματα εμπορίου κτλ καταψήφισαν ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας διευκρίνησαν οι εκπρόσωποι των χωρών αυτών ότι δεν έχουν αυτή την ίδια αντίληψη με μας για τα θέματα αυτά. Ήταν μια ενέργεια που δεν ήταν και πολύ φιλική απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξαν και άλλα ενδιαφέροντα θέματα που συζητήθηκαν Εν πάση περιπτώσει η αντιπροσωπεία ήταν ε, καλή, ενδιαφέρουσα, σωστά οργανωμένη και ήταν και ιδιαίτερα αθλητική γιατί τα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών είναι μοιρασμένα σε όλη την ε, Νέα Υόρκη και πηγαίναμε με τα πόδια από το ένα στο άλλο. Και δημιουργήθηκε μια νέα λέξη στα αγγλικά, ίσως αυτοί που ήταν στο στρατό τη γνωρίζουν, ήταν η, η πορεία θα έλεγα του αποσπάσματος της αντιπροσωπείας όλη την ημέρα εκεί. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Κρίμα που δεν έχουμε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε τα, τις ε, αποστολής αυτής. Η κυρία Λοχπίλερ. Δεν θα προσθέσω πολλά στα όσα είπε ο κ. Λάιχτφριντ. Διεξαγάγαμε συνάντηση με, τον, με την Μισελ Μπασελιέ, πρώην πρόεδρο της Χιλής, που τώρα ηγείται της ε, μονάδας αυτής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των γυναικών και που έχουν ανάγκη από χρηματοδότηση. Ήταν σωστό που ακούσαμε για θέματα για της κατάστασης των γυναικών σε περιόδους και ε, τόπους πολεμικών σειράξεων. Το δεύτερο που είπε είναι ότι θα ρίξει ιδιαίτερο βάρος στον στόχο της χιλιετίας ε, των ε, θανάτων γυναικών κατά τη διάρκεια του τοκετού και σε θέματα φτώχειας των γυναικών. Ήταν λοιπόν ιδιαίτερα ενθαρρυντική συζήτηση μαζί της και μάλιστα προσφέρθηκε να έλθει και στο Κοινοβούλιο την επόμενη φορά που θα επισκεφθεί τις Βρυξέλλες για να συνομιλήσει μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ εσείς κυρία Άλβινσον. Βέβαια είναι λίγος ο χρόνος που μένει. Σας ευχαριστώ πάντως ήθελα να σας ενημερώσω για το τι προέκυψε από την συζήτηση αυτή μέχρι τώρα 65η αυτή δηλαδή ε, συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα 65 ε, ψηφίσματα που ανταποκρίνονται σε υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θα σας πω όλες αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά δεν πιστεύω 6,5 ώρα πια ε, βραδινό Δευτέρας να τα ακούσετε όλα αυτά. Πάντως ε, ε, ενεκρίθησαν με συνένεση αυτά τα θέματα που βρήκαν απήχηση περισσότερο στα μέσα μαζική ενημέρωση ήταν αυτά που δεν έτυχαν συνένεση. Ιράν, Μιανμάρ, Βόρεια Κορέα, Μέση Ανατολή. Αυτά κυρίως ήταν τα θέματα. Συνολικά 11 ψηφίσματα της ε, ε, συνέλευσης. Βέβαια, στην πραγματικότητα δεν είναι καινούργια πράγματα αυτά, δεν ήταν πραγματικά νέα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα θεματικά ψηφίσματα, εξοδικαστικές εκτελέσεις, που καταδικάστηκαν βέβαια απανταχού, αλλά δόθηκε ιδιαίτερο βάρος σε θέματα που έχουν σχέση με τις ερωτικές προτιμήσεις των καταδικασμένων που είναι και ένα καυτό θέμα τώρα για την Γενική Συνέλευση και όπου οι απεσταλμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έθεσαν ιδιαίτερα το θέμα της, ε, του ευάλωτου των προσώπων ε, αυτών. Αυτό όμως αρχικά, το κείμενο αυτό αρχικώς αφαιρέθηκε, λόγω όμως δυναμικής παρεμβάσεως των Ηνωμένων Πολιτειών τελικά δέχθηκε η ε, πλειοψηφία. Το άλλο θέμα για την θανατική ποινή τώρα μια όλο και μεγαλύτερη ε, πλειοψηφία τάσεται υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής. Αυτό είναι σημαντική επιτυχία. Υπήρξαν και άλλα αμφιλεγόμενα ψηφίσματα σχετικά με ρατσισμό και θέματα ανεξιθρησκείας, αλλά βασικά ε, τήρησε σαφή γραμμή η Γενική Συνέλευση για τα θέματα αυτά. Νέοι κανόνες για την μεταχείριση γυναικών κρατουμένων. Αυτοί οι νέοι κανόνες δεν θα πρέπει να λησμονηθούν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς προχωρεί στην ανάληψη πρωτοβουλειών και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράδειγμα για την τέταρτη οδηγία για τα δικαιώματα των κρατουμένων και θα γίνει και μια παγκόσμια διάσκεψη το 2014 για τα δικαιώματα των ηθαγενών πληθυσμών. Αυτά είναι με λίγα λόγια, βεβαίως προσπαθώ να είμαι σύντομη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία μου. για την πολύ σύντομη αυτή σάρωση του ορίζοντα της 65ης ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον ο τρόπο με τον οποίο το επιτύχατε να είστε τόσο σύντομοι. Και τις επόμενες εβδομάδε θα συζητηθεί η σύνθεση αντιπροσωπείας ε, που θα μεταβεί στη Γενέβη. Υπάρχουν οκτώ διάφορα. Εδώ ε, επιθυμεί η κυρία Βεργιά να λάβει το λόγο. Στην αρχή της συνεδρίασης πήγα να το ρωτήσω, αλλά δεν έγινε αντιληπτή από την πρόεδρο. Τέλος πάντων είχαμε πολλά θέματα. Να προσπαθήσουμε να βρούμε το χρόνο για να συζητήσουμε τα της Τινησίας. Ε, σας έχω κουράσει για τη συνέχεια. Ζητώ τα ίδια. Όμως έγιναν εκεί σοβαρά πράγματα. 20, 30, 50 είναι οι νεκροί και ίσως πρόκειται αυτός ο κατάλογος να μεγαλώσει όπως είναι κατά, κατάσταση ώρα, την ώρα στην Τινησία. Και επομένω η υποεπιτροπή θα πρέπει να ασχοληθεί. Τα είπε η Μπάρμπαρα, κυρία Σάκ επίσης. θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη, ούτως ώστε τελικά να γίνει συζήτηση σε ολομέλεια, ενώπιον του σώματος. Αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό. Όμως, πέραν αυτού, αυτό δεν πάει να πει ότι δεν θα πρέπει που η Επιτροπή μας να το συζητήσει. Και να προβληματιστούμε, να το σκεφτούμε. Ακόμα και αν πλέον δεν μπορώ να πάω με την αποστολή στην Τινησία. Όπως προαναφέρθηκε, έχουμε δύο μέτρα δύο σταθμά εδώ. Ε, είχαμε κάποιους εδώ της πλειοψηφίας που αρνήθηκαν να εγκρίνουν τη συμμετοχή μου. Δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να πάω εκεί για να μάθω τι γίνεται. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με διαφορετικό τρόπο με την κατάσταση. Τέλος. Το τελευταίο θέλω να σας αναφέρω Μισό στον να βρω το σχετικό σημείωμα. κυρία Αρνό, είπε προηγουμένω ότι η εκπρόσωπο τύπου τη κυρία ε, Άστον ήταν κρυστάλλινη για τα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο. Να σας πω τι είπε. Απίθυνη έκκληση προς τις αρχές της χώρας να μην καταφεύγουν σε χρήση βίας. Τι είναι αυτό, ξεκάθαρη, ξεκάθαρη τοποθέτηση ενώ έχουμε 30 με 50 ε, θανάτους. Ούτε καν καταδίκασε αυτούς τους θανάτους. Απίστευτο αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταδίκη της βίας. Μα αυτά δεν είναι ξεκάθαρα. Αυτά είναι ανεπαρκή και ουσιαστικά σκανδαλώδη. Τι να πούμε. Έχουν συνηθίσει να υποφέρουν στην Τινησία. Δεν είναι καν αυτό. Πήγαν να διαμαρτυρηθούν, τους σκοτώσαν στον δρόμο και τα πτώματά τους τα πετάνε από εδώ και από εκεί σε όλη τη χώρα. Και καθόμαστε εδώ τώρα και συστάμε αμπελοφιλοσοφίζουν γιατί όλα αυτά τα τρομερά στη χώρα. Είναι ευθύνη όλων. Να καταδικάσει τα όσα γίνονται εκεί, είναι θέμα αξιοπιστίας της Ένωσης και του Κοινοβουλίου. Δεν θα πρέπει έτσι, χωρίς αντίδραση, να συνεχιστούν, να γίνουν όλα αυτά σε Ολομέλεια και στην Επιτροπή μας. Να δούμε τι γίνεται με αυτή τη δήλωση. Νομίζω ότι αυτά τα οποία είπε είναι ανεπαρκή ευχαριστώ. E, e, Έχετε Θα πρέπει αυτό να συζητηθεί και στην Ολομέλεια μας. Νομίζω θα να συζητήσουμε στο μέλλον. και στο διαβεβαιωμένο Προεδρείο. Όχι τι είπατε για την εκπρόσωπο τύπου και θα πρέπει πάντως να δεχθούμε ότι ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακά όσα έγιναν ε, κατά τις γιορτές όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία τα συζητήσαμε κατά το πρώτο σημείο μας. Όλες αυτές τις παραδιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλα όσα έγιναν Δίκη Χοντροκόφσκι, Λευκορωσία. Και για τους υποψήφιους, αλλά και για μέλη της αντιπολίτευσης. και το θέμα της τυνησίας. Δεν ξέρω, είναι τυχαίο ότι αυτά όλα γίνανε στις ε, διακοπές ή μήπω γίνανε επειδή σε αυτή την περίοδο δεν μπορεί το Κοινοβούλιο να αντιδράσει σε τέτοια πράγματα. Euronest, είχαμε τις συνεδρίαση. Τα διάφορα βήματα συνεννόησης. Η θα πρέπει να συζητήσει για την Λευκορωσία. Να ληφθεί κάποια απόφαση. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε τις αναβολές. Νομίζω θα υπάρξει ευκαιρία να γίνει διάλογος. Πάντως, έχει λήξει όμως τις οπότε θα πρέπει να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας. Κύριε Λόχμπιλε, θέλετε το λόγο. συμφωνώ. Θα πρέπει να ζητηθεί το θέμα της χώρας. Και κυρίως να γυρίσει η αποστολή. Κάτι τώρα για τους συνεργάτες μας, τη γραμματεία. Δεν ξέρω, πέστε μου αν ισχύει κάτι τώρα. Διάβασα στο EU Observer ότι η ψηλή χώρα όπως κάθε Άστον ευθυγραμμίζεται με το εμπάργο για την μη πώληση όπλων στην Κίνα. Αυτό το εμπάργο όπλων είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε από την Μέν. Είναι όλο αυτή η ιστορία. Να δούμε σε ποιες περιπτώσει δεν θα, θα αυτό το εμπάργο. Αυτό είναι μια ολόκληρη συζήτηση, αλλά για πέστε μου. Πότε θα συζητηθεί αυτό, γιατί είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν ξέρω, εκτός βέβαια, για να θεωρήσουμε ότι είναι αναλυθείτε αυτό που γράφει Small meeting, even if the public are maybe watching it to extent which we underestimate at our peril. That is an extremely good. Πάρα πολύ εύστοχα τα είπατε. Αφορά και θέματα θεσμικά. Πέμπτη και Παρασκευή συνδρίασε μέσα Δεκεμβρίου το Συμβούλιο. συζητήθηκε εκεί πέρα. Ε, σχέση με, με ε, τις πολιτείες, Κίνα, Ρωσία. Και συζητήθηκε για το περίπλοκο θέμα της άρσης του εμπάργου. Είναι περίπλοκο, δεν είναι θέμα μόνο ψηφίσματος. Επομένως, σας παραπέμπω στον κύριο Αλμπερτίνη όταν συνδυάσει η Επιτροπή Αφέτη. Θα κοιτάξουμε και εμείς από τη γραμματεία, μπορούμε να βρούμε τα σχετικά έγγραφα, από ό,τι βέβαια ξέρω. Όλα αυτά δεν είναι δημόσια. Τα έχω δει. Αλλά ό,τι και να προσφέρει κανείς για την ώρα του εμπάργου, υπάρχει εδώ και θέμα θεσμικό. Πώς περνάει κάτι από την υψηλή πρόσωπο και το κοινοβούλιο δεν παίρνει μυρωδιά. Σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε. Εξάντληση με τη μέση διάταξη. Και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ όλους και τους διερμηνείς, διότι μας επέτρεψαν να παρατηρούμε τη συνεδρίαση και να μας συμπαθάνε.